Καλημέρα συνάδελφοι, είναι παρούσα η συγγήτριά μας, οπότε ας είμαστε ακριβείς και σεβαστούμε και εκείνους που ήρθαν στην ώρα τους σήμερα το πρωί και ξεκινήσουμε την συνάντησή μας. Η κυρία Γιατεμάκη, επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας ε, ε, παρατηρήσεων των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήγε σε μια αποστολή με αυτό το σκοπό την παρακολούθηση των εκλογών στις 7 Νοεμβρίου στο Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ την προσωπία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για την παρακολούθηση των εκλογών. Έγιναν παρατηρήσεις και όσον αφορά, παρόλο που ήταν ειρηνικές οι εκλογές και η αντιπολίτευση μπορούσε να συμμετάσχει σε εκλογές, Συνολικά όμως οι εκλογές Δεν θεώρησαν οι παρατηρητέ ότι έγινε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό του Αζερβαϊτζάν λόγω των εκλογών που διεξήχθησαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θα αφήσω τις λεπτομέρειες ε, στην εισηγήτριά μα. Η κυρία λοιπόν Γιάννη Τενμάκη έχει το λόγο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, προσωπικό του Κοινοβουλίου, καλημέρα σε όλους, είναι ωραίο πρωινό. Και τα καλύτερα μέλη της Επιτροπής μας είναι εδώ. Ας μπω λοιπόν στο θέμα όμως. Ήμασταν 7 μέλη στην αντιπροσωπεία, συν το προσωπικό μας, 15 νομίζω σύνολο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τη δυνατότητα που μου δίνει να παρουσιάσω τις αρχικές παρατηρήσεις μετά την αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν και όπως είπε και ο Πρόεδρος τα πάντα ήταν ήρεμα και ειρηνικά. Αυτό ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό σημείο αυτό. Όμως, όμως, παρόλα αυτά, θα ήθελα να τονίσω αλλά δεν έγιναν όλα όπως έπρεπε. Η σωστή διεξαγωγή ε, των εκλογών δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει τα πάντα για, την, ε, για τον εκδημοκρατισμό της χώρας και για ομαλές εξελίξεις. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήγε σε διάφορες ε, περιοχές της χώρας καθώς και στο Βακού και πολλά μέλη είπαν ότι η γενική ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη και από πλευρά τεχνική η διεξαγωγή των εκλογών ήταν καλή. Όμω υπήρξαν σοβαρέ ελλείψει όσον αφορά τη διαφάνεια της ψηφοφορία ε, την προετοιμασία ε, των εκλογών, τους πίνακες, του εκλογικού καταλόγους κλπ. Οι εκλογές στο Αζερβαϊτζάν δεν οδήγησαν σε κάποια πολιτική συζήτηση και δεν ενδιαφέρθηκε και ιδιαίτερα ο λαός. Με τα βίας παρατηρήθηκε ότι διεξήγονται εκλογές. Σαν μην γινόταν εκλογές καθόλου. δεν υπήρχαν αφήσει. Δεν έγινε προκλητική εκστατεία ουσιαστικά. Δεν βγήκαν λόγοι. ούτε θεωρητικά υπήρχε η δυνατότητα να εκλεγεί διαφορετική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Μόνο 38 υποψήφοι της αντιπολίτευσης είχαν εγγραφεί στο Κοινοβούλιο που έχει 125 έδρες. και δεν ήταν ανεξάρτητη αναφορά στα μέσα ενημέρωσης. Οι ψηφοφόροι είχαν περιορισμένη πρόσβαση στις διάφορες ε, απόψεις και αμερόληπτη ενημέρωση και πληροφορίες για να μπορέσουν να κάνουν την επιλογή τους. Δεν έγινε δημόσια συζήτηση μεταξύ του κόμματος της πλειοψηφίας και των υποψηφίων της αντιπολίτευσης. Υπήρξαν πολλοί τετράλεπτοι μονόλογοι στην τηλεόραση. Δεν έγινε όμως ζωντανή συζήτηση με θέμα ένα πολιτικό πρόγραμμα για τη χώρα και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τα διάφορα κόμματα η αντιπροσωπεία μας, τα μέλη της αντιπροσωπείας μας προσπάθησαν επανειλημμένα να ρωτήσουν τους προέδρους των διαφόρων κομμάτων της αντιπολιτεύσεως να πούν ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Όμως δεν μπορούσαν να πούν τίποτα. Κατηγορούσαν μόνο το κόμμα της πλειοψηφίας και εκεί σταματούσαν. Τίποτα άλλο. μετά τις εκλογές, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες, καταλήξαμε σε τελική δήλωση για τα παρασκευαστικά τα αρχικά ε, πορίσματα και για την κοινοβουλευτική συνοδεύση του Συμβουλίου της Ευρώπης και για το γραφείο του ΑΣΕΙ, για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα πορίσματα θα τα βρείτε στους, στο φάκελό μας. Επιτρέψτε μου όμως να προβώ σε κάποια πολιτικά σχόλια. Σχόλια που βασίζονται στις παρατηρήσεις μας. Οι εκλογές και οι δημοκρατικές εξελίξεις στο Ζερβαϊτζάν πρέπει να ειδωθούν στο σωστό ε, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο. Δεν είναι η κατάσταση ίδια όπως εδώ στο κέντρο της Ευρώπης. Πάντα ήταν διαφορετική κατάσταση εκεί. δεν υπάρχουν ε, βαθιές ρίζες όσον αφορά τι δημοκρατικέ εκλογές στο Ιράν, ο Βόρειο Κάφκασο, η Αρμενία, η δημοκρατία τη Ρωσική Ομοσπονδία, η Γεωργία. Αυτοί είναι γείτονε του Αζερμπαϊτζάν. Και δεν ξέρουμε και ποια κατάσταση επικρατεί εκεί. Υπάρχει σαφής απάθεια στους ψηφοφόρους. Ίσως και στην Ευρώπη να ισχύει αυτό, αλλά εκεί είναι πολύ ορατή αυτή η απάθεια. Ακόμα και αν η επίσημη συμμετοχή ήταν πάνω το 50%. Υπήρχε έλλειψη ενδιαφέροντος όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές εκλογές και αυτό διότι η χώρα έχει προεδρικό σύστημα κυβέρνησης. Το κοινοβούλιο έχει ελάχιστες εξουσίες. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για την μη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου διεξήχθησαν οι εκλογές. Έχει πολύ δρόμο μπροστά της αυτή η χώρα μέχρι ότου να γίνει μια δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία της με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν, να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Εμπόριο και άλλα θέματα μέσω της συνεργασίας με τη χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εμπόριο νομίζω ότι είναι κοινό ζήτημα που αφορά και τις δύο πλευρές, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι βασικά αυτά τα θέματα που ε, ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά έχω να πω και καλώ τους συναδέλφους που είναι εδώ να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους και είμαι έτοιμη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να σας πω περισσότερα πράγματα για τις παρατηρήσεις μας και είμαι έτοιμη επίσης να ακούσω και κάποιες προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτριά μας. Ήταν πολύ εμπεριστατωμένη και ακριβής η παρουσίαση. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να μιλήσει, ο συνάδελφος ο κύριος Λίζα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την κυρία Μάκη γιατί ήταν εξαντλητικές οι πληροφορίες που μας έδωσε. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας και τη θέση των χωρών που παρακολούθησαν τις ε, εκλογές στο Αζερμπαϊτζάν ή τις ε, διάφορες οργανώσεις που παρακολούθησαν τις εκλογές στο, στο Αζερβαϊτζάν. Για παράδειγμα, η Αμερικανική κυβέρνηση είπε ότι σε καμία περίπτωση οι εκλογές δεν τήρησαν τις δημοκρατικές προδιαγραφές. Υπάρχει, υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των διεθνών παρατηρητών ενώ η αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής, ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κατέληξε διαφορετικό συμπέρασμα. Δεν υπήρχε συμφωνία σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των παρατηρητών εκλογών στο Αζερβαϊτζάν. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η διάσταση απόψε. Ε, Καλώς δεν βλέπω να ζητάει άλλο το λόγο. Κάποιος συνάδελφος θα θέλει να μιλήσει, οπότε να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για την απάντηση που ζητά ο κύριος Λίζε και για δεχόμενα σχόλια, τελικά σχόλια όσον αφορά την εργασία της. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και θα ήθελα να τη σχολιάσω μόνο και να πω ότι Εξαρτάται το πώς βλέπει και το άτομο τη δημοκρατία. Είναι προσωπικό θέμα. Υπάρχουν διαφορετικά ανοίγματα. Και όπως το είπα αυτό, όπως το ανέφερα και όταν συζητήσαμε με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΑΣΕ, οι διαπραγματεύσεις ε, δεν ήταν πάντα εύκολες διότι εμείς η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και οι εμπειρογνώμονες και εκείνοι που έχουν μείνει καιρό στη χώρα είχαν πολύ σοβαρές παρατηρήσεις όσον αφορά τις εκλογές, ότι δεν ήταν δημοκρατικές και δίκαιες. προσπαθήσαμε στην αντιπροσωπεία μας να ακολουθήσουμε τη μέση οδό. Να κατανοήσουμε την ιστορία, το πλαίσιο και ότι η δημοκρατία θα έπρεπε να είναι στόχος του Αζερμπαϊτζάν. Κάποιος θεώρησε ότι ήταν βήμα εκλογές προς τα πίσω. Κάποιοι είπαν ότι ήταν ε, βήμα πρόοδο εκλογέ. Και έπρεπε να καταλήξουμε σε μια κοινή δήλωση και δεν είναι πάντα τόσο εύκολο κάτι τέτοιο. Η ατμόσφαιρα όμως ήταν καλή και μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομερείς μας παρατηρήσεις στο φάκελο. Ευχαριστώ κυρία Γιάννη Τεμάκη. Εν τω μεταξύ ήρθε και ο Σβάγκελ ο οποίος θα κλείσει και τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, Θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με τα συμπεράσματά σας και τα όσα είπατε για τις εκλογές στην Ουκρανία, στο Αζερβαϊτζάν. Αλλά ήσασταν σε προνομιούχα θέση, ήσασταν παρόντες εκείνη την εποχή ακόμα και αν επικρατούσε κάποια απάθεια στον πληθυσμό όπως είπατε κάποια από τα ζητήματα δεν συζητήθηκαν. Δεν είχατε επαφές εσείς με τους υποψηφίους. Θα μπορούσατε να μας πείτε ίσως ποια είναι αυτά τα θέματα. Εκτός από την υποστήριξη του Προέδρου και του κόμματός τους. Δεν υπάρχουν άλλα πολιτικά ζητήματα κοινωνικής πολιτικής που να σημειώσατε ως κάτι που αποσχολεί τον κόσμο. Ιδιαίτερα θα με ενδιαφέρει να μάθω ότι λένε για τη λεγόμενη ευρωπαϊκή προοπτική του Αζερμπαϊτζάν. Προς τα πού έχει στραφεί και κατευθύνεται η χώρα, το μέλλον της, πού το βλέπει. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε σε αυτά. Ευχαριστώ. Ε, Κύριος Κάτσιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι, το Αζερμπαϊτζάν είναι ιδιαίτερη χώρα και είναι κρίμα να εκλέγεται ο πρόεδρος με λιγότερο από 90% υποστήριξη. Σε ρωτάνε, Αλή, είχες τη δυνατότητα να συζητήσεις με τους υποψήφιους της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές. Τι περιμένουν από τη θέση τους, από το ρόλο τους. Τι μπορούν να κάνουν. Μπορούν να επηρεάσουν τις μελλοντικέ εξελίξεις προς τον εκδημοκρατισμό του κράτους. Ευχαριστώ κύριε Κάτσιν. Λοιπόν, να, για να κλείσουμε, το λόγο τον έχει η κυρία Γιατενμάκη. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την πολιτική συζήτηση μεταξύ των διαφόρων κομμάτων, δεν διεξήχθη τέτοια συζήτηση. Ακόμα και αν ρωτήσουμε επανειλημμένα τα διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποια είναι η γραμμή σας για την κοινωνική πολιτική. Δεν μας δώσαν κάποια απάντηση, γιατί δεν υπάρχει. Δεν συζητείτε το θέμα, δεν υπάρχουν προγράμματα όπως έχουμε εμείς στις χώρες μας. Ήταν ενδιαφέρον αυτό που είδαμε και για μας. Και δεν ήταν μόνο ένας ή δύο που έθεσε το ερώτημα των πολιτικών προγραμμάτων. Όλοι, όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας μας το ρώτησαν και άλλες αντιπροσωπείες. Τους ρώτησαν. Ρώτησαν πολλές ερωτήσεις όσον αφορά τα προγράμματα. Κυρίως κοινωνικά πολιτικά ζητήματα. Και τους ρωτήσαμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα που συζητούν με το λαό. Αν υπήρξε, δεν υπήρξε προκριτική εκστρατεία. Βασικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούσαν την πλειοψηφία και αντιστρόφως, ανταλλαγή κατηγοριών γινόταν. Και ίσως και το Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν και ένα ζήτημα που συζητήθηκε. Δεν το είπαν ξεκάθαρα, αλλά όταν το συζητήσαμε με κάποιους μας είπαν ότι αυτό είναι το ζήτημα. που είναι ένα κοινό θέμα που απασχολεί τα κόμματα. Τώρα όσον αφορά την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματα των κομμάτων. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Όμως, συναντήσαμε και τον Πρόεδρο και υπουργού και διάφορους αξιωματούχους και σε αυτές τις συναντήσεις έλεγαν πάντα ότι θέλουν να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συνεχιστεί λοιπόν και να βαθυθεί η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Αζερβαϊτζάν. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται πολύ, πραγματικά ενδιαφέρονται για τη συνεργασία αυτή. Συνεργασία στον τομέα του εμπορίου. Ελπίζω όμως να είναι έτοιμοι να συζητήσουν και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων το θέσαμε το ζήτημα στον Πρόεδρο επανειλημμένα και στο μέλλον τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία θα είναι τα βασικά θέματα, ελπίζω, που θα τεθούν από την πλευρά μας, γιατί και υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα και τα κενά. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές, μόνο πριν τις εκλογές. Όταν όμως συναντήσαμε, κάποιους μετά τις εκλογές και μετά την δική μας επίσημη έκθεση δεν ήταν δύσκολο να συνεχιστούν οι συζητήσεις μαζί τους. Τους είπα παραδείγματος χάρη έτσι ευθέως ότι ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να συντάξουμε την έκθεσή μας, διότι γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι σήμερα ακόμα δεν ε, υπάρχουν δημοκρατικές εκλογές. Ίσως στο μέλλον να υπάρξουν. Να σας δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα για τις ομιλίες για την προεκλογική εκστρατεία αυτή που ήταν. Ένα παράδειγμα. Κυριακή, ημέρα εκλογών. Πήγαμε και εγώ πήγα σε πολλά εκλογικά τμήματα. Στο πανεπιστήμιο ήταν, στην περιοχή του πανεπιστημίου ήταν το πρώτο εκλογικό τμήμα. Ήταν πολλοί νέοι που παρατηρούσαν τις εκλογές. Και όταν πήγα τους ρώτησα από ποια κόμματα και μου είπαν ότι είμαστε από διαφορετικά κόμματα. Πήγα μετά στον κόσμο και τους ρωτούσα έναν έναν από ποιο κόμμα, σε ποιο κόμμα ανήκετε και όλοι ήταν από την πλειοψηφία εκτός από μια κυρία. Επειδή ήταν νέοι, άρχισαν να συζητούν τη δημοκρατία. Με ρώτησαν, εγώ προσπάθησα να τους πω τι σημαίνει να είναι κανείς στην αντιπολίτευση, τι σημαίνει να είναι κανείς στην κυβέρνηση. Λίγο πάνω από 20 ήταν νέοι, ήταν, τους ενδιέφερε πάρα πολύ το θέμα και τους ρώτησα μετά. Είδατε κάποιους λόγους, κάποια προεκλογική εκστρατεία, είδατε στο περιβάλλον σας κάποια κίνηση, στο περιβάλλον σας στη χώρα. Τι εκστρατεία υπήρξε. Και μου απάντησαν ότι δεν έγινε καμία τέτοια προεκλογική εκστρατεία και τους ρώτησα γιατί. Και μόνο μία κυρία, αυτή η κυρία, που ήταν από την αντιπολίτευση, μάλλον ανεξάρτητη, είπε ότι ήταν ανεξάρτητη. Αυτή απάντησε και είπε λόγω φόβου δεν έγινε εκστρατεία. Αλλά να πω κάτι άλλο. Στην, στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο συζητάμε τη συμφωνία σύνδεσης, το πακέτο, είμαι συγγήτρια για το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα ήταν πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτές τις εκλογές και αυτά που συνέβησαν, όλα αυτά θα συζητήσουμε στην Ολομέλεια. Όχι την επόμενη εβδομάδα, αλλά το Δεκέμβριο. Διότι ίσως θα ήταν καλό κάτι τέτοιο για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την ε, Συμφωνία Σύνδεσης. Λοιπόν, Ζητώ από τον κύριο Πρόεδρο να το θέσει αυτό το θέμα στη μέση διάταξη. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη Μάκη. Μπορούμε σίγουρα να λάβουμε υπόψη την πρότασή σας, όμως πιστεύω από πλευράς οργανωτικής ότι θα ήταν περίπλοκο κάτι τέτοιο, διότι το Δεκέμβριο η εργασία της Ολομέλειας, η μερίσια της Ολομέλειας ήδη έχει καθοριστεί, οπότε το να θέσουμε ένα θέμα που δεν έχει προβλεφθεί. Νομίζω ότι οργανωτικά είναι κάτι δύσκολο, όμως θα το θέσουμε το ζήτημα. πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκθεση του Πάουελ Ρόμπερτ Κόουαλ επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ουκρανίας σχετικά με τις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 31 Οκτωβρίου του 2010 και τη 15η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας που έλαβε χώρα, στο, πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο 4 και 5 Νοεμβρίου του 2010. Η έκθεση όσον αφορά λοιπόν τις τοπικές εκλογές στην Ουκρανία μπορεί να θεωρηθεί ένα, μια δοκιμή, ένα τεστ δημοκρατίας στη χώρα αυτή. Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρακολούθησε την εξαγωγή των εκλογών. Οι, οι πρόεδροι αποφάσισαν να στείλουν κάποιους συναδέλφους της Επιτροπής Συνεργασίας να πάνε στην Ουκρανία και να παρακολουθήσουν αυτή τη δραστηριότητα. Καλωσορίζω λοιπόν την πρόεδρο της Επιτροπής και τον κύριο Κοσλόφσκι που παρακολούθησαν ε, προσεκτικά την όλη αυτή διαδικασία. Α, δεν είναι εδώ. <laughs> λοιπόν, ε, τα ανέφερα λίγο πιο πριν, οπότε έπρεπε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόουαλ και μετά θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις πριν να δώσω το λόγο συναδέλφου να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριο κύριος λοιπόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, η αποστολή μου ήταν ε, ασυνήθιστη και ε, συγκεντρώσαμε την προσοχή και εξαιτία αυτού του γεγονότο, επειδή βρεθήκαμε στο επίκεντρο τη προσοχή, υπήρξε και κάποια μεγαλύτερη ένταση και άγχος. Θα ήθελα να σα πω ότι ε, Είχα μοιράσει το πρώτο ανεπίσημο έγγραφο και σήμερα είναι η δεύτερη εκδοχή της έκθεσης ε, για την αποστολή στην Ουκρανία με τα στοιχεία από τα εκλογικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να πω κάτι που είναι θεμελιώδες και δημιουργεί κάποιες μερικές φορές ε, ε, παρεξηγήσεις σε ό,τι αφορά την παρουσία μας στην Ουκρανία. Γιατί οι εκλογές αυτές δεν τήρησαν τις προδιαγραφές και τους κανόνες της ΟΑΣΕ. Δηλαδή, καμία οργάνωση, κανένα από του θεσμού που συνήθω παρατηρούν εκλογέ, ούτε το Συμβούλιο τη Ευρώπη, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η ΟΑΣΕ, ούτε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, έστειλαν επίσημα κανονικέ ε, αποστολέ παρατήρηση ε, εκλογών. Ούτε σε προκαταρκτική φάση, ούτε σε φάση παρατήρησης εκλογών. Οπότε, σε ό,τι αφορά την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για, την, για τις εκλογές αυτές υπάρχουν κάποια προβλήματα ως προς το τεχνικό στοιχείο. Φυσικά υπάρχει και το πολιτικό στοιχείο που θα το αναλύσω πιο διεξοδικά, αλλά αυτό θα ήθελα να τονίσω, γιατί παρόλο που μίλησα πολύ και έγραψα πολλά για το θέμα αυτό, δημιουργείται μερικές φορές ε, μια συνεννοησία ως προς το αντικείμενο της αποστολής. Βέβαια παρόμοιες αποστολές ε, είχε και η ΟΑΣΕ. Για παράδειγμα είχαμε συναντήσεις με πολιτικούς, με εμπειρογνώμονες, με άλλους παρατηρητές και αυτά τα ανέλησα διεξοδικά στην έκθεση για την αποστολή στην Ουκρανία και φυσικά στη συνέχεια είχαμε την, την συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας που έλαβε χώρα αμέσως μετά τις εκλογές και αυτή η αποστολή παρατήρησης των εκλογών κράτησε αρκετά, ένα οκταήμερο, γιατί αναλαμβάνω ακολούθησε η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας και αυτή η σχετικά μακροχρόνια παραμονή μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε πιο εμπεριστατωμένα αποτελέσματα. Και αμέσως μετά την επιστροφή, γιατί γύρισε στις 6 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία, αμέσως μετά την επιστροφή μου, ήδη από τις 11 ε, Νοεμβρίου κατήρτισα το πρώτο σχέδιο της έκθεσης και είπα και στον κύριο Μπρόκ και στον κύριο Γκάλερ ότι ένα τρι, τριήμερο κράτησαν ουσιαστικά οι εργασίες εκπόνησης αυτής της έκθεσης. Πιο σύντομα δεν γινόταν, γιατί στην Ουκρανία δεν μείναμε μέχρι την Τρίτη, αλλά μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Οπότε είχα μόνο ένα τριήμερο ουσιαστικά για να προετοιμάσω την έκθεσή μου από τις εκλογές. Ήταν πολύ σημαντικό και έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό στην έκθεσή μου να περιλάβω όλα τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν, δηλαδή όλη την αλληλογραφία μου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας ή και την αλληλογραφία που είχα με εκπροσώπους ε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά τα θέματα, όλες αυτές οι επιστολές έχουν και πολιτικό χαρακτήρα και σας επιτρέπουν να εξάγετε και εσείς συμπεράσματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο μηχανισμό παρατήρηση εκλογών, αλλά εδώ έχουμε περισσότερο μία άντληση πολιτικών συμπερασμάτων και αυτό ήταν ενδιαφέρον για την Ουκρανία. Γι' αυτό και επισύναψε όλες αυτές τις επιστολές, γιατί έτσι εξηγούνται και τα προβλήματα που ανέκυψαν στη διάρκεια των εκλογών και στο πλαίσιο των εκλογών. Υπάρχει το θέμα της ελευθερίας έκφρασης, το θέμα των συχνοτήτων για μέσα μαζικής ενημέρωσης και το θέμα του διαδικτύου. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα και όλα αυτά τα πορίσματα και των, εκλογών, των διαφόρων αποστολών παρατήρηση τα έλαβα στην έκθεση, προκειμένου να καταλήξω στο συμπέρασμα αυτό. Είχαμε την οργάνωση ΟΠΟΡΑ και μια άλλη οργάνωση που έχουν τις μεγαλύτερες εμπειρίες και τις πιο πλούσιες εμπειρίες από την παρατήρηση εκλογών στην Ουκρανία και επίσης ε, είχα τακτικές επαφές με την Κεντρική ε, Επιτροπή Εκλογών στην Ουκρανία που επίσης ήταν ο οργανισμός αναφοράς. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, σας παραπέμπω φυσικά και στο έγγραφο που συνέταξα και θα ήθελα να πω ότι οι εκλογές, οι τοπικές, οι δημοτικές εκλογές στην Ουκρανία δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε με τις βουλευτικές εκλογές ούτε με τις προεδρικές εκλογές. Και υπάρχει κάποια σύγχυση γιατί οι προεδρικές και οι βουλευτικές εκλογές κατά τη γενική γνώμη των παρατηρητών των τελευταίων χρόνων αλλά και τη, με βάση τη δική μου γνώμη γιατί ήμουνα στους δύο γύρους των τελευταίων προεδρικών εκλογών έγιναν με βάση τις ε, δημοκρατικές προδιαγραφές. Στηρίθηκαν σε μεγάλο επίπεδο οι δημοκρατικές προδιαγραφές για εξωκοινωτικές χώρες. Φυσικά δεν συγκρινώ με τις κοινωτικές χώρες. Και αυτό το λέω μετά από πολυετή εμπειρία που είχα σε αποστολές παρατήρησης εκλογών στην ΟΑΣΕ πριν να γίνω Ευρωβουλευτής. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε τις εκλογές της αυτοδιοίκησης με τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές ούτε μπορεί να θεωρηθεί η Λιδία της δημοκρατικότητας του συστήματος. Γιατί από αυτή την άποψη θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε πολιτικά συμπεράσματα που είναι πιο επικριτικά απέναντι στην Ουκρανία σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές. Για παράδειγμα, είχαμε έναν δρυμή πολιτικό αγώνα γύρω από τις εκλογές και όχι μόνο αγώνα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αλλά και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αντιπροσωπεία της ε, Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ήρθαμε σε επαφή με πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, του Αρσένιο, Αρσένη Γιατσένιο για παράδειγμα, που είναι πολύ μικρότερο σε από το κόμμα της ε, Γιούλιας Τιμοσέγκο και μετά το πέρα των εκλογών ε, ασκήσαμε κάποιες επικρίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών και η θέση του Γιατσένιουκ ήταν σχετικά μετριοπαθής παρόλο που ο ίδιος είναι κόμμα αντιπολίτευσης σε σχέση με το κυβερνόν κόμμα. Πάντως ε, υπάρχει ε, ένα σύστημα δημοκρατικό, προχωρά η διαδικασία εκδημοκρατισμού και φάνηκε αυτό περισσότερο από τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές. Πάντως ήταν δυσανάλογο το ενδιαφέρον ε, των πολιτών εξαιτία της μικρής αρμοδιότητας που έχουν οι δήμοι και οι κοινότητες. Η αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία δεν είναι αυτοδιοίκηση με μεγάλες εξουσίες όπως έχουμε στην Πολωνία, στη Γερμανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό οι εκλογές έχουν περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα. Από ουσιαστική άποψη δεν είναι λίδια λίθος της δημοκρατίας γιατί δεν έχουν σημαντικές αρμοδιότητες. Δεν υπάρχει ουσιαστική αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια ανάλυση με βάση τους μηχανισμούς που έχουμε και κυρίως ε, να κάνουμε κάποια πολιτικά, κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Εγώ είχα αρκετά επικρίσεις για τις ε, τοπικές εκλογές. Δεύτερη φορά στην ιστορία το, της Ουκρανίας άλλαξε ο εκλογικός νόμος πολύ λίγο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο τα αποτελέσματα των εκλογών αλλά και η, η ποιότητα του εκλογικού νόμου εκτός του ότι τελευταία στιγμή λίγο πριν τις εκλογές εγκρίθηκε αυτός ο εκλογικός νόμος είχαν συνέπειες και στην διεξαγωγή των εκλογών και στην ουσία πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν σε εκλογές σε κάποιες επαρχίες της Ουκρανίας εδώ δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε γενικευμένα συμπεράσματα γιατί δεν έχουμε μηχανισμό. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή να αποτιμήσουμε τις εκλογές σε κάθε όμπλαστ, σε κάθε επαρχία δηλαδή της Ουκρανίας. Αλλά από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε μπορούμε να επισημάνουμε κάποια φαινόμενα ανησυχητικά. Για παράδειγμα στο Λβόβ και στο Κίεβο, το κόμμα πατρίδα της Γιούλια Τιμοσέγκο, το κόμμα Μπατκεφτσίνα, δεν μπόρεσε στην ουσία να λάβει μέρος στις εκλογές. Παρόλο που οι δύο αυτές επαρχίες είναι επαρχίες όπου η Γιούλια Τιμοσέγκο έχει αρκετή εκλογική δύναμη. Και αυτό τη της τη της ε, τοπική επιτροπή, εκλογικής επιτροπή. Στην πράξη λοιπόν, ο νέος εκλογικός νόμος οδήγησε σε αρκετά προβλήματα γιατί δόθηκε ευκαιρία στι τοπικέ εκλογέ να κάνουν ερμηνεία αυτού του εκλογικού νόμου με αποτέλεσμα να αποκλειστούν ορισμένα κόμματα από την ε, ουσιαστική συμμετοχή στι εκλογέ σε ορισμένε επαρχίε. Δεν μπορούμε επίση ε, να ε, εκτιμήσουμε την επιλογή αυτών των ελαττωμάτων του νόμου στο συνολικό αποτέλεσμα των εκλογών. Έγιναν κάποιες δημοσκοπήσεις και είδαμε και τα exit polls σε σχέση με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Αλλά εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε μηχανισμό αντίστοιχο με τη ΣΟΑΣΕ για να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. Και αυτή τη φορά η ΟΑΣΕ δεν παρακολούθησε τι εκλογέ στην Ουκρανία. Πάντω οι λεπτομέρειες ε, θα τις βρείτε στην έκθεσή μου. Μπορούμε να καταλήξουμε σε τρία συμπεράσματα. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση της ε, αυτοδιοίκησης είναι σημαντικό θέμα. Να μην επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα του εκλογικού νόμου, αλλά μια και η Ουκρανία είναι μια χώρα που έχει ενταξιακή προοπτική, θα πρέπει να προβεί σε κάποιες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Οι διοικητικές αυτές μεταρρυθμίσεις ε, συμπεριλαμβανομένων και των μεταρρυθμίσεων της αυτοδιοίκησης είναι θεμελιώδες ζήτημα για την Ουκρανία και θα πρέπει να προχωρήσει. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής συνεργασία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και απέστειλα σχετική επιστολή στον πρόεδρο με τις παρατηρήσεις μου. Εμείς ε, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ασχοληθήκαμε κυρίως με το θέμα της συνεργασίας ε, για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στην Ουκρανία. Κάτι άλλο που προέκυψε από τις εκλογές είναι ότι χρειαζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα θεσμικό όργανο που μονίμως θα βρίσκεται στην Ουκρανία και θα είναι σε θέση να προβαίνει σε σωστή εκτίμηση των εκλογών. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είχαμε στη, στη διάθεσή μας ένα κατάλληλο μηχανισμό για να προβούμε σε διεξοδική και πλήρη αξιολόγηση των εκλογών αυτών στην Ουκρανία. Και τα συμπεράσματα των, ε, της παρατήρησης των εκλογών δεν συμπεριλήθηκαν στο τελικό έγγραφο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας και αυτό γιατί δεν καταλήξαμε σε... δεν υπήρχε μια ενιαία θέση των εκπροσώπων της ε, Ουκρανίας. Υπήρξε αντιπαράθεση των διαφόρων πολιτικών κομμάτων της Ουκρανίας, γι' αυτό υπήρξε διαφωνία, υπήρχε τέτοιος διχασμός στην Ουκρανική αντιπροσωπεία ως προς την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των εκλογών που αποφασίσαμε τελικά τα συμπεράσματα για την παρατήρηση των εκλογών ή για τα αποτελέσματα των εκλογών να μην τις συμπεριλάβουμε στο τελικό έγγραφο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κόβουαλ για την αξιέπαινη εργασία σας. Όλοι την εκτιμούμε και πραγματικά θα τη θεωρούσαμε ένα καλό θέμα για συζήτηση. Όμως πρέπει να επιτρέψω τον εαυτό μου με την τόρμη που με χαρακτηρίζει σε αυτή τη φάση να αναφερθώ στα διαδικαστικά. Δηλαδή, στο πώς διαβιβάζεται αυτή η εξέπαινη εργασία σας στην ύπατη εκπρόσωπο και περιέχει και κάποιες ε, προτάσεις η έκθεσή σας. Και είναι εξωτερικός φορέας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν προφανώς συνδεδεμένος, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια ομάδα εκλογικού συντονισμού στην οποία συμπροεδρεύω, μαζί με τον κύριο Ζολή και έχει σαν σκοπό να αξιολογεί τις διαδικαστικές πτυχές της εκλογικής διαδικασίας και θέματα πολιτικά με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή μας. Λοιπόν, υπενθυμίζω τον κανονισμό. Προ, από το πρεζίντερε, το λατινικό προστατεύω βγαίνει η λέξη πρεζιντέντε, πρόεδρος. και οι συστάσεις και οι παρατηρήσεις οδήποτε συναδέλφου πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοβούλιο και μετά στα εξωτερικά, στους εξωτερικούς φορείς. Στην αξιέπαινη εργασία σας εσείς κάνετε μια πρόταση. Τη δημιουργία μιας υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως παρατηρήσεων όλων των ειδών των εκλογών των χωρών της γειτονίας και αυτό προφανώς είναι αξιοσέβαστη σκέψη σας, αλλά δεν μπορεί να είναι άποψη όλου του Κοινοβουλίου αν αυτό δεν έχει συζητηθεί, όπως ήδη είπα, ε, στα διάφορου φορεί του σώματο που προβλέπετε, δηλαδή στην ομάδα εκλογικού συντονισμού και την Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων. Ο κύριο Μπροκ έχει ζητήσει το λόγο και του απευθύνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα να μιλήσω πρώτο εγώ τώρα, ε, γιατί καθυστέρησα. Θέλω να μιλήσω άλλοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση αυτή. Γιατί με κάνει να συνειδητοποιήσω μερικά πράγματα και να καταλάβω ότι και εμείς ε, μπορούμε να κρίνουμε και να κρινόμαστε με βάση τις ίδιες μας αρχές. Κατά τη διάρκεια των εκλογών πιστεύω δεν υπήρξαν τίποτα φοβερές ε, παραβιάσεις αλλά στην προετοιμασία των εκλογών υπήρχαν προβλήματα. Και αυτό αναγράφεται σε δύο προτάσεις μόνο στο σημείο 3-4, δηλαδή διαδικαστικά τεχνάσματα που απέκλεισαν το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στα εκλογικά του κάστρα. Δεν κατάφεραν υποψήφοι του κόμματος αυτού να κατέβουν με το όνομα του κόμματο. γιατί το σφετερίστηκαν κάποιοι άλλοι και κατέβηκαν με αυτό το όνομα στις εκλογές ο συνδυασμό. Άρα δεν είναι ανεξάρτητη η εκλογική διαδικασία και αδιάβλητη και δεν μπόρεσε να αλλάξει η παραμονή των εκλογών. Στο ε, Λβόβ και στο Κίεβο που είπαμε ότι είναι κάστρα τη αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να κατέβει αντιπολίτευση γιατί κατεβαίνει άλλο συνδυασμό με το ίδιο τη το όνομα. Μα πριν αρχίσουν καν οι εκλογέ, αυτό είναι νοθεία των εκλογών, δεν είναι. Και αυτό θα πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα και να το τονίζουμε και όχι σε μια υποπαράγραφο και να το κρύβουμε πίσω από τέτοιες τυπικές ε, προτάσεις. Το λέτε στην έκθεσή σας κύριε Κόβαλα, τι λέτε ότι δεν μπόρεσαν να καταγραφούν ε, ως ε, αυτός εκλογικός συνδυασμός και ήρθε η κυρία Τιμοσέκο και είπε ότι μποϊκοτάρει τις εκλογές. Μα δεν μπορούσε να μποϊκοτάρει, δεν μπορούσε να συμμετέχει σε εκλογές γιατί τις είχαν πάρει το όνομα του συνδυασμού και είχαν κατέβει κάποιοι άλλοι, λες, και ήταν ελεύθερη της απόφαση αυτό. Περίεργο μου φαίνεται αυτό ως διατύπωση εδώ. Επίσης γνωρίζετε ότι Παίζει ρόλο και η σειρά των υποψηφίων σε ένα ψηφοδέλτιο και πάντα και η σειρά των ψηφοδελτιών ορίζεται ανεξάρτητα. Δεν είναι κατά σειρά εμφανίσεως όποιος ήρθε πρώτος και ε, καταγράφεται. Και το εκάστοτε περιφερειακό κόμμα πάει και γράφεται πρώτο και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτό είναι δεύτερη νοθεία. μπορούμε να συζητήσουμε και το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και το σύνταγμα ε, της ε, Πορτοκαλί Επανάστασης. Φρόντισε και ο επικεφαλής ε, των μυστικών υπηρεσιών που είναι στο συνταγματικό δικαστήριο να αλλάξουν τέσσερις δικαστές του συνταγματικού δικαστηρίου και να έχει διαφορετικό σχετισμό και να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύνταγμα. Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα, δεν είναι. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών ασφαλεία. μπορεί να έχει λόγο στην επιλογή των δικαστών. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή υπάρχει διάκριση των εξουσιών εδώ, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Έχουμε προβλήματα. Καταλαβαίνω από την άλλη βέβαια ότι έφερε σταθερότητα η νέα κυβέρνηση, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν καν σε θέση να πράξει ούτε αυτό. Και γι' αυτό ε, είχαν και αυτά τα αποτελέσματα στις εκλογές. Και λόγω αυτής της σταθερότητας αποφάσισαν και η κυβέρνηση και η Βουλή προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση για τους λόγους που σας ανέφερα απέτυχε να το πράξει αυτό. Εξού και η κριτική μου προς την εκλογική αυτή διαδικασία. Και το συμπέρασμα δεν είναι ότι πρέπει να επιδεινώσουμε εμεί θέσει μας τώρα και τις σχέσεις με την Ουκρανία. Όχι. Ζώνη ελευθερών συναλλαγών και συμφωνία σύνδεσης πρέπει να προχωρήσουν και η διευκόλυνση ε, χορήγηση σε διαβατηρίων. Έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν ζητώ εδώ επιβράδυση των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία λόγω των εκλογών. Το αντίθετο, μάλιστα. Πάντως, ε, και θέλω να το πω, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κρινόμαστε και με τα κριτήρια που επιβάλλουμε ε, και σε κάποιους άλλους. Είναι προειδοποιητική αυτή ε, η στάση. Αφήστε που άμα πάτε να μιλήσετε με μέλη της κυβέρνησης δεν τα αμφισβητούν ούτε τα ε, διαψεύδουν. Σου λένε την άλλη φορά δεν θα ξαναγίνει. Ωραία. Ε, λοιπόν, αφού και οι ίδιοι τα παραδέχονται, θα συζητάμε και να μην δίνουμε την εντύπωση ότι στη μεγαλοψυχία μα και στη μεγαλοθυμία μα τα παραβλέπουμε και πάμε παρακάτω. Γιατί θα έχουμε πουτινοποίηση και της Ουκρανίας. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα προβλήματα με την Ουκρανία. Αυτό είναι χρέος μας. Να κάνουμε και τέτοιες αξιολογήσεις ειλικρινείς και με όλες τις χώρες με τις οποίες ε, συναλλασσόμαστε. Όχι με καλοπισμούς και με ρετουσάρισμα να καμουφλάρουμε τα προβλήματα. Αυτά. Και κύριε Κόβαλ, εμείς έχουμε κάποιες αξίες δημοκρατικές, κράτους δικαίου και προσπαθούμε να δώσουμε ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στην Ουκρανία. Και δεν θα βοηθήσουμε με κάποιες τρευλές ερμηνείες. Ε, είναι παράδεκτο αυτό. Αφήστε που αποθαρρύνει και τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Τα πάντα αλλάζουν. Είναι ρευστά. Αντί για κοινοβουλευτισμό μπορεί να επανέλθει και το προεδρικό σύστημα. Εντάξει, αυτό εναπόκειται σε κάθε χώρα είναι ελεύθερη Βούλη των πολιτών, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζονται εξή δύο. Πρώτον, η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει ευκαιρία ε, ε, δίκαιη και ίση να γίνει η πλειοψηφία και επίσης θα πρέπει να έχουμε διάκριση των εξουσιών. Άλλο πράγμα εκτελεστική και άλλο πράγμα η δικαστική εξουσία. Αυτό σημαίνει για μένα κράτος δικαίου και δημοκρατία. Και στην προετοιμασία των εκλογών είχαμε αυτή την κατάσταση που ενδεχομένως να διακύβευε ε, αυτά που σας λέω. Πότε ήταν εκλογέ δεν θυμάμαι, το 2007 ε, οι βουλευτικές, που ήταν δίκες και ε, ανοιχτές και έντιμες. Τώρα δεν θα πρέπει να ζητούμε για να αλλάξει το, ο εκλογικός νόμος για να γίνει τύπου αυτοδιοικητικών εκλογών που έγινε τελευταία στιγμή και παρά την ε, συμβουλή και την υπόδειξη της ε, Επιτροπής της Βενετίας. Που δεν την άκουσαν, αλλά έκαναν αυτό που νόμιζαν. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η χώρα αυτή. Έχουμε κοινή πορεία, θέλουμε κοινή εξέλιξη, αλλά ε, με όρους κράτους δικαίου, επαναλαμβάνω, και δημοκρατίας. Και να το ξεκαθαρίσουμε. Για τη δική μας Επιτροπή είχε δεσμευτεί πάρα πολύ, αγωνίστηκε για την Πορτοκαλή Επανάσταση. Δεν θα πρέπει να τα εμπομολήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Μίρσκι, ο επόμενος. Αν μπορείτε να είστε πιο σύντομος, διότι βλέπω ότι μας περνάει η ώρα. Κύριε Ζούσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και διάβασα και πολύ προσεκτικά την έκθεση ε, για τις εκλογές στην Ουκρανία. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, οι συνάδελφοι πήγαν στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των εκλογών, έτσι, τρεις μέρες μόνο έμειναν εκεί. Και είμαι βέβαιος ότι δεν είχαν πολύ χρόνο ε, για να ακούσουν και να ε, αξιολογήσουν την κατάσταση και πολιτικά. Ε, από τη Λετωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρωσία, Σερβία, Ηνωμένε Πολιτείε πήγα και εγώ με 12 συναδέλφου, εκπροσώπου Δήμων και κοινοτήτων. Ήμασταν επίσημοι εκπρόσωποι τη οργάνωση Δήμων και κοινοτήτων. Και Πήγαμε στη ε, Σεβαστούπολη, στο Ντονιέτ, στη Βίνιτσα και σε άλλες πόλεις. Και ακολουθήσαμε ε, λοιπόν αυτή την πορεία και ε, βγάλαμε τα εξή συμπεράσματα. Είναι νεόκοπη κυβέρνηση στην Ουκρανία και δεν έχει μεγάλη εμπειρία, αλλά συνολικά οι εκλογές μπορούν να θεωρηθούν δημοκρατικές. Δεν διαπιστώσαμε μεγάλα σφάλματα για προβλήματα που να μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Χαιρόμαστε που η κυβέρνηση της Ουκρανίας θέλει στο μέλλον να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και ε, να ε, προσαρμόσει τη χώρα. Θέλω να τονίσω επίσης και να υπογραμμίσω ότι μπορούμε να αυξήσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να βοηθήσουμε την κυβέρνηση της Ουκρανίας να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Ακριβώς ε, έτσι ώστε ο νόμος αυτός να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνει η Ουκρανία ένα πόσπαστο τμήμα της Ευρώπης που είναι και να αισθάνεται και έτσι όμως. Τώρα, τρεις μέρες μόνο τόσο μικρός αριθμός πολιτών να πηγαίνει σε μια χώρα 50 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων δεν έχει αρκετό χρόνο για να διαπιστώσει τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόβαλ για την έκθεσή του, για την άποψή του ε, που είναι αρκετά ισορροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μίρσκι. Ο κύριος Γκάλερ για δύο λεπτά αν μπορείτε. Ένα λεπτό διαδικαστικό παρακαλώ. Ωραία. Σας δίνουμε το λόγο. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, λύπη που δεν άκουσε την ε, εισαγωγή μου ο κύριος Μπροκ και αυτό θα ήθελα να μου δώσετε το λόγο όσο είναι για να μπορέσω να τον απαντήσω. Να το απαντήσω. Θέλετε να μιλήσετε πριν το τέλος της συζητήσεως? Αμέσως τώρα? μετά τις παρατηρήσεις του κυρίου Μπροκ. Θα ήθελα φυσικά να απαντήσω στον κύριο Μπροκ. Γι' αυτό αν παραμείνει στην αίθουσα να περιμένω, αλλά δεν θέλω να φύγει πριν να ακούσει την απάντησή μου. Καλώς. Ο κύριος Γκάλερ για δύο λεπτά έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, δύο λεπτά δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Ας ξεκινήσω. Λοιπόν, μια εισαγωγική παρατήρηση. Όντως, Τελευταία στιγμή μας κάλεσε η κυβέρνηση, γι' αυτό δεν μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε τον παραδοσιακό μηχανισμό που έχουμε για την παρατήρηση των εκλογών. Αν είχαμε απορρίψει αυτό το αίτημα όμως θα ήταν και πρόφαση της κυβέρνησης να πει ότι τους καλέσαμε και δεν ήρθανε, γιατί δεν ενδιαφέρονται. Εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, αποτέλεσμα κλασικού τύπου και φυσιολογικής παρατήρησης εκλογών. Και για τα συμπεράσματα πρέπει να πω ότι δεν τα θεωρώ στην πλειοψηφία τους αντικειμενικά και εύστοχα. Στη συνέχεια, Επιτροπή συνεργασία κοινοβουλευτική στις 4 και 5 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση δεν έγινε κανείς λόγος για τις εκλογές αυτές. Τρίτον, ούτε δημοκρατικές ήταν οι εκλογές ούτε δίκαιες. Δεν ξέρω ο συνάδελφος εδώ ε, τι γνώμονα και τι κριτήρια έχει. Μήπως του είπε αυτά ο ε, επικεφαλής της ε, Υπηρεσίας Ασφαλείας στο πολυτελές εστιατόριο των Βρυξελών μεζών του Σίνι, του Σίνι ε, και στο δείπνο που είχαν οι δυο τους. η οργάνωση Οπόρα και κάποιοι άλλοι έκαναν λόγο για μη δημοκρατικές εκλογές και συμφωνώ και εγώ. Τώρα, ε, έρχομαι στην ίδια την έκθεση, σελίδα 7. Το εκλογικό σύστημα, χωρίς καμία κριτική, παρουσιάζεται και, ε, όπως έχει. Μα ε, από τη δομή την ίδια είναι αμφισβητούμενο, είναι αμφιλεγόμενο, κυριαρχεί ένα κόμμα και όλα τα άλλα είναι κατακαιρματισμένα και με το πλειοψηφικό σύστημα που έχουν κιόλας είναι πολύ μονομερή η σύνθεση των οργάνων για των αποτελεσμάτων. Η έκθεση λέει απλώς ότι δεν έγιναν εκλογέ στο Κίβεβο. Ήταν τακτικισμός αυτός γιατί καταργήθηκε εκεί το, ε, ε, καταργήθηκαν κάποια συνοικιακά συμβούλια ε, επίτηδες για να νοθευτούν οι εκλογές. Ε, γίνεται λόγος και για τις εφορευτικές επιτροπές αλλά δεν ε, ε, γίνεται λόγος για τη σύνθεσή της ε, εκάστοτε εφορευτικής επιτροπής γιατί κατά πλειοψηφία επευλήθη εκεί και στη σύνθεση των μελών και ποσοτικά το κυβερνών κόμμα. Τώρα, για τις αρχές του εκλογικού νόμου απλώς περιγράφεται αυτός, δεν αξιολογείται και στο σημείο 34 τα είπε και ο κύριος Μπροκ ε, γίνεται λόγος για μποϊκότ. Τι μποϊκότ, αφού δεν είχε δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Μποϊκότ είναι αυτό. Ε, δίνεται λάθος εντύπωση. Ορισμένοι, λέει, από τους ε, υποψηφίους ε, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της προκλήσης εξαρτίας, άρα δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν. Και ωραία, τι είναι αυτή η δήλωση τώρα, παρηγοριά στον άρρωστο τους πιάσανε και δεν μπόρεσαν να κατέβουν σε εκλογές. Μπράβο. Μπόρεσαν τελικά. Α, μπόρεσαν. Δηλαδή του συνέλαβαν και μετά του άφησαν ελεύθερου και μπόρεσαν να συμμετέχουν σε εκλογέ. Ωραία παρηγοριά είναι αυτή. Ε, συμπεράσματα. Ε, και πάλι δεν συμφωνώ με τα συμπεράσματα. Δεν είναι αντικειμενικά. Πρώτο συμπέρασμα. Είχε κάποια στάνταρ, είχε κάποια πρότυπα και προδιαγραφές πετύχει η Ουκρανία, τώρα τα έχει εγκαταλείψει. Και δεν είναι και καλή η σύσταση ε, της συνολικής αναθεώρησης του εκλογικού συστήματος. Η αναλογική ε, απεδείχθη ε, καλό σύστημα στι προηγούμενε εκλογές και συμφωνούν όλοι ότι ήταν ε, τα αποτελέσματα και η συμμετοχή των κομμάτων σωστή και ελεύθερη Οπότε δεν νομίζω ότι στι κοινοβουλευτικέ εκλογέ χρειάζεται τώρα να θυγεί, να αναθεωρηθεί ε, ο εκλογικό νόμο και να χρησιμοποιηθεί ο νόμο που ισχύει για τι αυτοδιοικητικέ και δημοτικέ εκλογέ. Άλλο που λέει η έκθεση. Οποιαδήποτε υποχώρηση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών θα ήταν ανεπιθύμητη. Μα αυτό συμβαίνει ήδη. Οπότε Και πάλι ωραιοποιείται την κατάσταση. Τέλος. Πώς να το πω, δεν ξέρω και πώς να τα διατυπώσω. Η δήλωση της κεντρικής κυβέρνησης να αλλάξει τον εκλογικό νόμο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και με ελπίδα. Ναι, εντάξει, η ελπίδα δεν είναι κριτήριο άσκηση πολιτική κανονικά. Δεν θα έπρεπε να λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά να λέμε ξεκάθαρα τι είναι οι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ και τι κάνει η Ουκρανία και πρέπει να τηρεί και πώ θα κρίνεται η Ουκρανία και αυτή. Και επίση, δεν θα πρέπει να έχουμε διατυπώσει τύπου το Ωστόσο, οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ στην Ουκρανία, ε, παρόλο που γνώρισαν μεγάλη ε, διεθνή προβολή, ε, οι ε, τοπικές ε, και περιφερειακές αρχές δεν έχουν και μεγάλη εξουσία στη χώρα. Και τι σημαίνει αυτό. Α, ωραία, εντάξει. Είχε νοθεία στις εκλογές, δεν πειράζει. Σιγά την εξουσία που έχουν και αυτοί εκεί πέρα και τις δυνατότητες παρέμβασης. δεν είναι σκόπιμο να γράφουμε τέτοια πράγματα σε εκθέσεις μας. Όταν κάνουμε παρατήρηση εκλογών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή, απλώ να γραφεί στα πρακτικά. Γιατί αν ψηφίζαμε, εγώ θα ήμουν υποχρεωμένο να ζητήσω καταψήφιση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Δεν μείνατε στα δύο λεπτά, τα ξεπεράσατε κατά πολύ. Ο κύριος Τάνοκ θα τα καταφέρει. Κύριε Τάνοκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα επαναλάβω εγώ τα σχόλια που έκανα προηγουμένω. Καταρχήν, εγώ είμαι αντίθετο με το να είναι παρατηρητή στο κοινοβούλιο στι τοπικέ εκλογέ όπω και βασικέ στρατηγικέ χώρε όπω είναι η Ουκρανία. Δεν είμαστε τοπικοί βουλευτέ, πολιτικοί, όπω αναφέρθηκε η τοπική κυβέρνηση δεν έχει σημαντικέ εξουσίε εθνικέ και διεθνεί, έχουν σημαντικού πόρου βεβαίω και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά για να προβάλλουν το ρόλο των τοπικών πολιτικών βαρώνων για τα κόμματά του και επηρεάζουν τελικά και το εθνικό προσκήνιο. Δεν είναι δουλειά μας αυτή και παρακολουθώ και με ενδιαφέρει αυτό ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έστειλε εκπροσώπους από εθνικούς βουλευτές, έστειλαν από το Κογκρέσο από τα, των Περιφερειών από τη Βουλή των Περιφερειών. Αν μα δοθεί στο μέλλον τέτοια εντολή, να τη στείλουμε στην Επιτροπή των Περιφερειών την εντολή, που είναι ο αρμόδιος φορέας Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείται με τοπικέ και περιφερειακά θέματα, και να στείλουν λοιπόν ε, ε, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης να πάνε για να παρακολουθήσουν τοπικές εκλογές, περιφερειακές ε, εκλογές, γιατί παρατηρούμε σε όλο τον κόσμο τοπικές εκλογές. Και αυτό αένα συνέχεται. Ήταν η Γεωργία πριν, η Ουκρανία τώρα, δεύτερη φορά, μετά ξέρω εγώ. Τελικά θα περνάμε όλο μα τον καιρό κάνοντα παρατηρήσει εκλογών. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό σαν πολιτική πριν τελικά γίνει κάτι ανεξέλεγκτο. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο κύριο Γκάλερ, τα άκουσα η κατάσταση στην Ουκρανία δεν είναι τέλεια, αλλά ούτε θα είναι βλέποντα τα μέσα που υπάρχουν την παρακολούθηση των εκλογών. Δεν θα ξέρουμε ακριβώ τι έγινε. Είναι τεράστιο εγχείρημα οι τοπικέ εκλογέ. Χιλιάδε υποψήφοι. Πού να βγάλει κανεί άκρη. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα που να βγαλει κανει απαράδεκτα βέβαια. Είναι απλά τα πράγματα στη χώρα μα όσον αφορά το ψηφοδέλτιο. Και δεν είναι υποψηφίο άλλο. Ε, είναι αλφαβητική σειρά στο ψηφοδέλτιο, οπότε ξεπερνιέται το πρόβλημα. Ε, το να καταχωρούν τοπικές ε, αρχέ και να βάζουν πάνω στο ψηφοδέλτιο πάντα αυτού του παλιού που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους νέου υποψήφιους. Πάει αλφαβητικά το όνομα υποψηφίου και όχι τα κόμματα ε, στη χώρα μου. Δεν ξέρω. Ε, και είπα ότι το Μπιούτ δεν μπορούσε να συμμετάσχει σαν μπλοκ. Είμαστε, έχουμε συνασπισμό σε εθνικό επίπεδο στη χώρα μου και το Μπιούτ κινείται εντό τη Ράντα. Δεν έχουν όμω νομικό καθεστώ. Δεν είναι καταχωρημένο κόμμα. Το συντηρητικό κόμμα είναι και όχι η συμμαχία στη χώρα μου. Θα μπορούσε λοιπόν, δεν μπορούσε να είσαι υποψήφιος του συνασπισμού, ούτε σε τοπική ε, ε, ε, στι τοπικέ εκλογέ. Μπορεί κανεί να πει ότι είμαι συντηρητικό, αλλά μπαίνω τελικά στο εκλογικό κατάλογο, στο ψηφοδέλτιο των φιλελευθέρων. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να πα στο κόμμα τη Τιμοσέκο αν είσαι από το άλλο κόμμα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορούσαν να, μπουν στο κόμμα, να εγγραφούν σαν να ανήκουν στο κόμμα της Τιμοσέγκο. Ούτε και στο Μπακευσίνο, ούτε κανένας άλλος που εκπροσωπεί το, το Μπακευσίνα δεν μπορεί να, το, να, να συμμετάσχει με αυτόν τον τρόπο σαν να ανήκει σε συνασπισμό. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και από τα δικαστήρια. Εν γέννη είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κανεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, διότι είχαμε πάρα πολύ μικρή παρουσία, μόνο στο Κίεβο ήμασταν και κάπου αλλού. Και όταν έχεις τώρα 10.000 υποψηφίους κορπισμένους σε όλη τη χώρα και τόσες ε, τοπικές συνιστώσεις να κινούνται, πού να καταλάβεις αν είναι εκλογές. Δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτό, να μην ασχολούμαστε εμείς με την παρακολούθηση, με την παρατήρηση των τοπικών εκλογών. Κύριε Κέλαμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κόβαλ για την έκθεσή του και συμφωνώ βεβαίως με το συμπέρασμά του ότι η Ουκρανία χρειάζεται διοικητική μεταρρύθμιση πρώτα απ' όλα. Ωστόσο όμως Είμαι και εγώ λίγο μπερδεμένο ως προς το μήνυμα της έκθεσης αυτής. Ήταν ανησυχητικές οι εξελίξεις στην Ουκρανία. διότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έκλεισαν ε, πρόσωποι της αντιπολίτευσης ε, και υποψήφοι εμποδίστηκαν από το να συμμετέχουν στις εκλογές. Ήταν σαφές ότι οι μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν να παρεύουν στην εκλογική διαδικασία. Η ελευθερία της έκφρασης επίσης ε, ήταν αμφίβολη για να το πω έτσι και τελευταία στιγμή άλλαξε και ο εκλογικός νόμος. Με βάση όλα αυτά λοιπόν ε, ε, το συμπέρασμα που λέει ότι προχωράει όλο και περισσότερο η δημοκρατία και ο δημοκρατισμός της χώρας, αν το κατάλαβα καλά, μας οδηγεί σε κάποια σύγχυση. Εν πάση το συμπέρασμά σας είναι ότι ήταν μικρά μόνο τα επεισόδια και τα προβλήματα και γενικά οι εκλογές έγιναν με τρόπο ε, έτσι, ευπρεπή. Ε, και κάτι άλλο που με ενοχλεί κάπως και με οδηγεί σε ε, σύγχυση είναι ότι δεν φύγουμε αυτά τα προβλήματα. Ε, προσπαθούμε να κρατήσουμε αποστάσεις ή ακροθυγώς λίγο ε, να τα θίξουμε. Ακούσαμε τον συνάδελφο Χόκμαρκ στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα που είπε ότι επιστρέφει ο ίδιος από την Ουκρανία και πολλοί Ουκρανοί περιμένουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Όχι ότι κάνει τα στραβά μάτια και στρέφει το βλέμμα του από τα προβλήματα. Θέλουν να, θέλουν να βοηθήσει το Κοινοβούλιο την Ουκρανία να αντιμετωπίσει ε, τα προβλήματα με ε, ειλικρίνεια στην προσέγγιση του. Εγώ λοιπόν αμφιβάλλω ε, κατά πόσο η έκθεση αυτή μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση που θέλουν. Συμφωνώ απολύτω με τον συνάδελφο Έλμαρ Μπρόκ ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να φέρουμε πιο κοντά στην Ευρώπη την Ουκρανία, αλλά να έχουμε, μάλλον να επικρατούν ε, φυσιολογικές συνθήκες για την αντιπολίτευση, διάκριση των εξουσιών και ελευθεροτυπία, που ήταν ε, μέγα επίτευγμα της Πορτοκαλή Επανάστασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλαμ. Κύριος Λίζεκ, αν μπορείτε να τέσσετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ προσπαθώ να είμαι λακωνικός και μάλιστα να μην εξαντλήσω καν το δίλεπτο. Θα ήθελα να σας δώσω μία πληροφορία σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας. Στην πρώτη αποστολή που συμμετείχαν οι κύριοι Κόβαλ και Κοζουόφσκι. Θα ήθελα να πω στον κύριο Γκάλερ και στους ε, υπόλοιπους ότι στη διάρκεια των ε, συναντήσεων που είχαμε κατά την συνεδρίαση ε, της Επιτροπής Κοινοβουλευτική Συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Πρωθυπουργό Αζάροφ, με τον Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων και με τον Επικεφαλή των Μυστικών Υπηρεσιών που με βάση τις δικές μας προδιαγραφές και στάνταρ πραγματικά διαδραματίζει πολύ περίεργο ρόλο σε όλες αυτές τις συναντήσεις ε, διαβιβάσαμε τις ανησυχίες μας και νομίζω ήταν χειρό το μήνυμα που δώσαμε ότι οι προδιαγραφές αυτές δεν συνάδουν με τις ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή με τις προδιαγραφές ενός δημοκρατικού κράτους. Δεν ήταν ε, η αξιολόγηση των εκλογών τμήμα του επίσημου προγράμματος συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας, αλλά σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε με εκπροσώπους του κυβερνώντο κόμματο και τη ε, αντιπολίτευση ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Συναντηθήκαμε και με την κυρία Γιούλια Τιμοσέγκο, με τον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, με τον κύριο Ταράσουκ, με τον κύριο Γιατσένιουκ. Όλε αυτέ οι ανησυχίε, όλα αυτά τα αρνητικά μηνύματα και τι επικρίσει τι ε, διαβιβάσαμε και είχαμε και πολλά ιδρύματα και διεθνείς οργανώσεις που είχαν μεταφέρει αντίστοιχα αρνητικά σχόλια και εμείς τα μεταφέραμε και προς την κυβέρνηση και προς την αντιπολίτευση. Νομίζω ήταν πολύ χειρό το μήνυμα της αντιπροσωπείας μας προς τις πολιτικές δυνάμεις Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ και ο Λαντσμπέργκης έχει το λόγο. Αν μπορείτε δύο λεπτά ο Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής για τα συμπεράσματα και του ορισμού για την Ουκρανία που χρησιμοποιούνται. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα γενικό παρατηρητή. Δεν έχω την εντύπωση ότι ο εκδημοκρατισμό στην Ουκρανία προχωρεί όλο και περισσότερο. Το αντίθετο, θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους. Ε, και που λένε ότι ήταν τελείως μη δημοκρατικές εκλογές στην Ουκρανία. Τις εκλογές στη Ρωσία πώς τις ορίζετε. Μία και μόνη υποψηφιότητα ήταν για την εκλογή του Πρόεδρου. Και ο επόμενος Πρόεδρος ε, θα εκλεγεί από δύο, δύο εκλέκτορες. Θα συμφωνήσουν μεταξύ του. Αυτές τι εκλογές πώς τις αξιολογείτε. That friendly regime. Και ε, σε ό,τι αφορά τις φιλικές σχέσεις, το φιλικό καθεστώς είναι πιο φιλικό της Ουκρανίας ή της Ρωσίας, είναι καλύτερο της Ρωσίας. Πώς τα αξιολογείτε εσείς όλα αυτά τα θέματα. <clears throat> Καλώς ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Κύριε Κόουελ, εσείς για να ολοκληρώσετε. Ο κύριος Μπρόκ εγκαταλείπει την αίθουσα. Τον καλό να παραμείνει αν θέλει να ακούσει την απάντηση του εισηγητή. Εάν αποσιάσει θα διαβάσει τα πρακτικά. Κύριε Κόβολ, έχει το λόγο. Ε, ε. Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι ειλικρινά που φεύγει ε, από την αίθουσα ο κύριος Μπρό και δεν πρόλαβα, δεν τον πρόλαβα για να απαντήσω και να ακούσει την απάντησή μου. Ελπίζω ο κύριος Γκάλερ να του μεταφέρει τα σχόλιά μου. Η πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα καλά η μετάφραση του κειμένου του της έκθεσης δεν ήταν σωστή, γιατί ε, φαίνεται να υπήρξε παρεξήγηση. Εγώ συμφωνώ με τις εκτιμήσεις των κυρίων Μπρόκ και Γκάλερ σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Γιατί η Ουκρανία βρίσκεται ήδη στα μισά του δρόμου προς την ε, ευρωπαϊκή προοπτική και το κλίμα του, της συμπατκευσίνα της πατρίδας ε, είναι, ε, ανοίξει έναν συνασπισμό. Υπάρχει το και το, ή το κόμμα της Δυνατής Ουκρανίας ή της δικής μας Ουκρανίας είναι κόμματα φιλικά προς εμάς και πραγματικά είναι δύσκολο να καταλήγουμε σε τέτοια αρνητικά συμπεράσματα. Αλλά αυτό γίνεται αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές προδιαγραφές, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αλλά εγώ προσπαθώ να αποφύγω μονοσήμαντες πολιτικές δηλώσεις. Προσπαθώ, παρόλο που εγώ μπορεί να συμφωνώ με το ΕΛΚ στην εκτίμηση των εκλογών, προσπαθώ να καλύψω ένα ευρύτερο πολιτικό φάσμα γιατί είμαστε κοινοβουλευτική επιτροπή. Δεν μπορώ να προσποιούμε ότι ε, είχαμε πλήρη μηχανισμό παρατήρησης εκλογών όπως η ΟΑΣΕ και ότι μπορούμε να ε, εκπονούμε εμπεριστατωμένες εκθέσεις παρατήρησης εκλογών όπως αυτές της ΟΑΣΕ. Ήταν πολύ περιορισμένε οι δυνατότητέ μα. Μόνο πολιτική αξιολόγηση των εκλογών ήταν δυνατή. Παραλαμβάνω από τεχνική άποψη δεν είχαμε του μηχανισμού. Και δίκιο έχει ο κύριο Στάνακο ότι μπορεί να είναι λάθο αυτό το είδο παρατήρηση εκλογών, παρατήρηση και των δημοτικών εκλογών. Πάντω, το έγγραφό μου δεν είναι τόσο επίσημο. Και σίγουρα, αν έπρεπε να το εγκρίνουμε ως ε, έκθεση επιτροπής θα έπρεπε να είχαμε υιοθετήσει διαφορετικό, διαφορετική διαδικασία. Επαναλαμβάνω την το πρώτο σχέδιο του κειμένου το εκπώνησα μέσα σε τρεις μέρες. Συνήθως για εκθέσει είμαστε πολύ πιο σχολαστικοί, αλλά δεν είχαμε χρόνο για κάτι τέτοιο αυτή τη φορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες ε, παρατηρήσεις. Για τα σχόλια του κυρίου Αλμπερτίνη. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αλμπερτίνη. Όντω υπήρχε αυτό το στοιχείο τη ε, βιασύνη, της ε, ασάφειας ως προς το χαρακτήρα αυτού του εγγράφου. Αλλά θα ήθελα να σε ενημερώσω για τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε. Γι' αυτό και σα έκανα αυτή την εισαγωγή. Και συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις που έκανε ο πρόεδρό μα, ο κύριος Αλμπερτίνη, ό,τι αφορά τι ερωτήσει του κυρίου Μπροκ. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν προβλήματα με τη μετάφραση. Γιατί Νομίζω ότι το κείμενο ανταποκρίνεται σε αυτά που είχαμε πει και μεταξύ μας για την αξιολόγηση των εκλογών αλλά και τη δεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας. Σε ό,τι αφορά το... τη σειρά εμφάνιση των κομμάτων στα ψηφοδέλτια, όντως διαπίστωσα ότι υπήρξε μια προτίμηση και μια υπεροχή του κυβερνώντος κόμματος. Αλλά σε μια πολιτική έκθεση δεν μπορούμε να κάνουμε τεχνικέ αναλύσει για τον τρόπο διεξαγωγή εκλογών, όπω γίνεται συνήθω σε λεπτομεριακέ εκλογέ παρατήρηση. Αλλά δεν ήταν τέτοια αυτή η αποστολή παρατήρηση. Σε ό,τι αφορά την ε, ακύρωση τη αναθεώρηση του συντάγματο, αυτό δεν έχει σχέση με τι τελευταίε εκλογέ. Αλλά έχουμε πρόβλημα σχετικό στην Ουκρανία, γιατί πολλέ φορέ, μετά το 2004 όλα τα κόμματα και η αντιπολίτευση ήθελαν αλλαγή του συντάγματος του 2004, ακόμη και το κόμμα των επιτροπών, το κυβερνόν κόμμα. Αυτό μπορεί να το εκτιμήσει ο καθένα όπω θέλει. Πάντω όλα τα κόμματα και κυβερνών συνασπισμό και αντιπολίτευση ζήτησαν μετά το 2004 αλλαγή του συντάγματο. Επίση, ε, ήθελα να πω ότι εμεί δεν έχουμε μηχανισμό εκτίμηση εκλογών. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε μονολεκτικά αν ήταν δημοκρατικές ή αντιδημοκρατικές. Εγώ ρώτησα τη γνώμη και των ε, αρχηγών της αντιπολίτευσης. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε όμως μονολεκτικά ήταν όμω ορισμένες επαρχίες όντως υπήρξαν ατασταλίες. Έλαβαν χώρα πολλές, ε, πολλά προβλήματα. Σε πολλές επαρχίες ήταν κακή η οχι εκλογες σε ορισμένε επαρχιες οντως υπηρξαν ατασταλιε ελαβαν χωρα πολλες πολλα προβληματα σε πολλέ επαρχίε ηταν κακη η διεξαγωγη σε τρει-τέσσερι επαρχίε δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια τη αντιπολίτευση. Δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν κόμματα τη αντιπολίτευση. Από αυτή την άποψη, όντω δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τήρηση των δημοκρατικών προδιαγραφών και αυτό το είπα κατηγορηματικά. Ω προ αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία μεταξύ μα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί είχατε τόσο ε, έντονο τόνο. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση μεταξύ μα. Εγώ μίλησα για πολιτικά συμπεράσματα και σε αυτό συμφωνήσαμε. Δεν ήταν τεχνική αποστολή παρατήρηση. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε διεξοδική αποστολή παρατήρηση. Επίση, ε, κύριε Γκάλερ, γιατί ε, με ρωτήσατε στα συμπεράσματα τη Επιτροπή Κοινοβουλευτική Συνεργασία δεν αναφέρθηκαν οι εκλογέ. Αυτό δεν οφείλεται στη διαφωνία που υπήρξε στην κοινοβουλευτική πλευρά, στη δική μα πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σαφή και κατηγορηματική. Η Ουκρανική πλευρά δεν μπόρεσε να συμφωνήσει σε περιεχόμενο συμπερασμάτων. Οπότε δεν μπορέσαμε ούτε σε μια ελάχιστη συμφωνία να καταλήξουμε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να εξαιρέσουμε τελείως συμπεράσματα για τις εκλογές για να μην ε, κατηγορηθούμε ως υποκειμενικοί. Πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ενωμένο και ήταν πολύ ε, σωστό γιατί δείξαμε ότι η, Ευρωπαϊ... κοινοβουλευτική αντιπροσωπή και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι συσπηρωμένη και ενωμένη. Και αυτό φάνηκε στη στάση μα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτική Συνεργασία. Και αυτό θα φανεί στο ψήφισμα θα πρέπει να καταλήξουμε σε κοινή θέση για να έχει βάρος το πολιτικό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν υπάρχει διχασμός, διχασμός μεταξύ μας θα ερμηνευτεί πολύ αρνητικά αυτό το μήνυμα στην Ουκρανία γιατί η Ουκρανία ενδιαφέρεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολουθεί με πολύ προσοχή τα μηνύματα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης συμφωνώ απόλυτα με τα συμπεράσματα του κυρίου Γκάλερ. Θα ήθελα να επισημάνω μόνο το εξής για τον ε, κατάλογο των, ε, των κομμάτων και τη σειρά καταγραφής. Εγώ τον έφερα αυτό στην έκθεση. Αυτό ήταν σαφές ότι υπήρξαν ατασταλίες εκεί. Δεν ήταν πρόθεσή μου να τις ακρύψω. Επίσης το ίδιο σαφές είναι ότι ε, υπήρξε ελάχιστος χρόνος για την καταγραφή και αυτό ήταν πολύ αρνητικό. Όλα αυτά που είπατε για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής με βρίσκουν σύμφωνο. Επίσης και εγώ είπα ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει εξουσίες. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στις παραβιάσεις και στην εκλογική ατασταλία. Απλώς ζήτησα να θέσει η Ουκρανία την διοικητική μεταρρύθμιση ως προτεραιότητα. Γιατί οι Ουκρανοί πολίτες που συμμετέχουν στις εκλογές έχουν την αίσθηση ότι συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα που θα οδηγήσει σε αυξημένες αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης. Και αυτό δεν ισχύει στην Ουκρανία και αυτό διαταράσει κάπως τη δημοκρατική τάξη. Γιατί η δημοκρατική τάξη απαιτεί να δοθούν εχέγγυα στους πολίτες που συμμετέχουν σε εκλογές ότι η ψήφος τους έχει βάρος, έχει μία αξία, ότι δεν έχει μόνο τεχνικό χαρακτήρα, αλλά πραγματικά επηρεάζει το συσχετισμό των εξουσιών. Αυτό είναι σημαντικό. Γι αυτό, αυτό λέω στην έκθεση. Δεν θα ήθελα τα μηνύματά μας να ερμηνευτούν στην Ουκρανία ως εσωτερική αντιπαράθεση και διχασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, Τελικά ίσως έχει δίκιο ο κύριος Στάνοκ μετά από όλα αυτά, ότι πραγματικά δεν πρέπει να στέλνουμε αποστολή παρατήρηση στις δημοτικές εκλογές, εκτός και αν έχουμε έναν μηχανισμό που θα μας επιτρέπει να αξιολογούμε και από τεχνική άποψη αντικειμενικά τέτοιες τοπικές εκλογές, γιατί ίσως εκεί έγκυται το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Λίσεκ. Έχετε δίκιο και άκουσε ο κύριος Λίσεκ την θέση μας απέναντι στις Ουκρανικές αρχές. Το είπαμε προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις και στο κόμμα Σβόμποντα. Ε, είχαμε τον κύριο Σβόμποντα μάλλον από τους σοσιαλιστές στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπή. Είχαμε τον κύριο Λίσεκ. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι και μιλήσαμε με τις πολιτικές δυνάμεις. Πολλές φορές το λάθο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι δεν φαίνεται συσπηρωμένο και ενωμένο σε ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε μια ενότητα μεταξύ μα και μια συμφωνία. Κύριε Κέλαμ, εγώ δεν θα ήθελα να καταλήξω κάποια οριστικά πολιτικά συμπεράσματα, γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω εγώ στο όνομα ε, ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο στη δήλωση και στο ψήφισμα που θα εγκρίνουμε στο Στρασβούργο θα έχουμε ε, μια κάλυψη του πολιτικού φάσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και για να εκπονήσουμε αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Εγώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα στις εκλογέ. Κύριε Λαντσμπέργκη, σε όλε αυτέ τι πολιτικέ εκτιμήσει θα πρέπει και για το δικό μα κύρος, αλλά και για να προσπίσουμε την έγκλη και το κύρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να κρατήσουμε ένα, το αίσθημα του μέτρου. Όλε αυτέ οι παρατηρήσει δεν αλλάζουν το εξή γεγονός ότι για τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές ε, οι προδιαγραφές στην Ουκρανία είναι οι υψηλότερες δυνατές ό,τι αφορά τις ε, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Δεν μπορούμε όμως ε, να πιανόμαστε τις δημοτικές εκλογές που ήταν λιγότερο ήταν λιγότερο υψηλές οι προδιαγραφέ και να πούμε ότι η κατάσταση έχει μεταστραφεί και ότι ο εκδημοκρατισμός αναχαιτίστηκε. Νομίζω ότι η Ουκρανία έχει καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατικότητα των εκλογών. Δεν θα πρέπει με τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές να χάσει την καλή φήμη και την υπόλοιψη που έχει χτίσει η Ουκρανία για τη δημοκρατικότητα των εκλογών της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να είμαστε και εμείς αξιόπιστοι κύριε ε, για να μην δείξουμε ότι είμαστε πιο σε ό,τι αφορά την εκτίμηση εκλογών σε άλλε χώρε και αυτή τη φορά ε, στην, ε, στις δημοτικές εκλογές στην Ουκρανία ήμασταν πολύ πιο αυστηροί και ουσιαστικά ε, απαξιώνουμε ολόκληρη τη δημοκρατική μεταρρύθμιση τη Ουκρανίας που που την αναγνωρίσαμε. Μπορεί να μην έχει προχωρήσει με βάση τι τελευταίε εκλογέ στον εκδημοκρατισμό, αλλά ούτε έχει υποχωρήσει η Ουκρανία. Σα ευχαριστώ για όλε τι ε, παρατηρήσει. Θα πρέπει να κρατήσουμε αίσθηση του μέτρου, ισορροπία και ηρεμία και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να είμαστε ενιαίοι και να έχουμε ενωμένη φωνή στο ψήφισμά μας. Νομίζω ότι με κοινοβουλευτική ταπεινοφροσύνη και με τριοπάθεια άκουσα τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και με αυτό το πνεύμα ελπίζω να συνεργαστούμε και να συντάξουμε το ψήφισμα που θα είναι δίκαιο και αντικειμενικό όσο γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ όσοι συμμετείχα στη συζήτηση. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκάλερ για τις ε, επικρίσεις του, αν και πιστεύω ότι διέλυσε τις παρατηρήσεις, τις ανησυχίες ε, και τις αμφιβολίες. Κρίμα που έφυγε ο κύριος Μπρόκε δεν με άκουσε. Πάντως ε, οι διαφωνίες ε, που φάνηκαν εκ των προτέρων νομίζω ότι κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχουν μεταξύ μας. Ευχαριστώ κύριε Κόβαλ. Δυστυχώς που σας δώσω κύριε Μίνσκι το λόγο διότι έχουμε ένα κατεπήγον και ζητώ και να επιτρέψετε αλλαγή της ημερήσιας διάταξης αντί να ακούσουν τον κύριο, κύριο Μποντής να ακούσουμε τον κύριο Γκάλερ διότι πρέπει κάποιο να φύγει πιο γρήγορα. Ο αντιπρόεδρο μπορεί να φύγει πιο γρήγορα να αλλάξουμε τη σειρά. Αν συμφωνάτε, λοιπόν, πάμε στην σχέσει Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου πρώτα. Είναι μια έκθεση που ο κ. Λουίζη Ναρμπόντ επικεφαλής της ε, ε, αποστολής Τη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκή Ενώσεω στο Συμβούλιο Συνεργασία του Κόλπου στο Ριάντ, Μόνο εκπρόσωπο στην περιοχή και έχει ευθύνη για όλη την περιοχή. Λοιπόν, κύριε Μποντή, έχετε εσεί το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη συζήτηση που διεξάγεται όσον αφορά αυτή την έκθεση που αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και θα ήθελα να αναφερθώ στα διάφορα σημεία που είναι σήμερα οι σχέσεις μας λοιπόν και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εξελιχθούν στο μέλλον. Να πω πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα, να επενθυμίσω ποια είναι αυτή, αυτό το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Έξι χώρες ε, στην περιοχή του Κόλπου είναι το Κοβέιτ, το Μπαχρέιν που συμμετέχει, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Σουλτανάτο του Ομάν. Μοναρχικά καθεστώτα έχουν όλες αυτές οι χώρες και να επενθυμίσουμε ότι είναι ο μόνος οργανισμός με διαδικασία ολοκλήρωσης που ακολουθεί και στην περιοχή εκεί και στον αραβικό κόσμο γενικότερα. Προφανώς αυτό το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου που έχει μια στατηγική θέση μεγίστης σημασίας γιατί από τη μία πλευρά έχουμε τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου που είναι απέναντι από το Ιράν, είναι η αραβική ακτή ε, του κόλπου, του αραβικού και περσικού, ε, είναι γείτονα στο Ιράκ της Ιεμένης, στο Συμβούλιο του Κόλπου και είναι κοντά στη Σομαλία. Είναι σημαντικό το ειδικό φάρος διότι οι χώρες αυτές είναι πάνω, αντιπροσωπεύουν πάνω από ένα τέταρτο των χωρών που συμμετέχουν στον Αραβικό Σύνδεσμο. Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας παίζουν ρόλο διαμεσολαβητικό, όπως είναι η Αραβική Πρωτοβουλία για την Ειρήνευση που απορρέει από μια πρόταση του βασιλέως της Σαουδικής Αραβίας. Η κρίση του 2008 στο Λίβανο επελήθη κυρίως χάρη σε μια διαμεσολάβηση που ήταν πρωτοβουλία του Κατάρ οι χώρες του Συμβουλίου συνεργασία του Κόλπου είναι σημαντικές πολύ οικονομικά, διότι παράγουν και έχουν και αποθέματα φυσικού αερίου και έχουν υδρογονάνθρακες και να επενθυμίσω σχετικά με αυτό ότι οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου είναι οι πρώτοι προμηθευτές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες. Πολύ σημαντικός και ο ρόλος τους ο χρηματοπιστωτικός στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Τα, ε, τα, οι πόροι των χωρών αυτών, τα sovereign funds, είναι το 1 τρίτο του συνόλου των ε, πόρων αυτών στον κόσμο. Ε, πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Είμαστε σχεδόν στο νεκρό σημείο, θα μπορούσα να πω, 20 χρόνια διαπραγματευόμαστε για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, διαπραγματεύσεις που δεν κατέληξαν κάπου και δεν ολοκληρώθηκαν και είναι ρεκόρ αυτό. Είναι η πιο παλιά διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τρίτη χώρα, με τρίτο φορέ και που δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας έχει σαν στόχο να επαναπροωθήσει την όλη διαδικασία, να επενθυμίσει ότι η σύναψη στις Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών θα πρέπει να θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν στόχος με προτεραιότητα και να ζητήσουμε μια γρήγορη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ε, απ' την άλλη πλευρά θέτει και μια αρχή αυτή η έκθεση, δηλαδή ότι οι σχέσεις μας με τις χώρες συνεργασίας του κόλπου δεν θα πρέπει να τοποθετείται επί ενός εμπορικού επίπεδου και μόνο. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε μια σχέση πελάτου προμηθευτού στα πλαίσια αυτό των, ε, της, αυτής συμφωνίας ελευθερών συναλλαγών που δεν έχει συναυθεί ακόμα. Πηγαίνουμε πιο μακριά, προτείνουμε τη δημιουργία μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης σε πολιτικό και στατικικό επίπεδο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει περισσότερη, να είναι πιο ορατή στην περιοχή, κυρίως δίνοντας πιο σημαντικά μέσα, ε, να, είναι, να εκπροσωπείται καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και η εκπροσώπησή μας να βελτιωθεί. Ο κύριος Ναρμπόν την εξασφαλίζει μέχρι τώρα, τον οποίον θα μπορέσουμε να ακούσουμε και του υποβάλουμε ερωτήσεις αλλά θα κερδίσουμε εάν υπάρχει εκπροσώπηση ε, του ε, Συμβουλίου Συνεργασίας στον χώρο του κόλπου μάλλον στις πρωτεύουσες των χωρών να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και θέλουμε σε ύψιστο επίπεδο συζητήσεις με τακτικές συνόδους κορυφής με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τώρα έχουμε σε διπουργικό επίπεδο συναντήσεις και πολύ συχνά οι χώρες μας εκπροσωπούνται μόνο σε τεχνικό επίπεδο Υπάρχει περιθώριο για πολιτική συνεργασία. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενθαρρύνει αυτή τη διαδικασία της ολοκλήρωσης των χωρών ε, του Συμβουλίου Συνεργασίας ε, του Κόλπου. Ε, λοιπόν, υπάρχει, είναι αργή διαδικασία, αλλά υπάρχει και είναι η μόνη διαδικασία ολοκλήρωσης και στην περιοχή της συγκεκριμένη και στον αραβικό κόσμο. Και άρα μπορεί να ανταλλαγούν εμπειρίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης και χωρών συνεργασίας του κόλπου. Υπάρχουν πολλά διπλωματικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια. Έχουμε το Ιράν, κίνδυνος ε, εξοπλισμών στην περιοχή. Η σταθεροποίηση του Ιράκ είναι ένα άλλο θέμα. η κατάσταση που κρατεί στην Ιεμένη, άλλο θέμα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη Σομαλία. Δηλαδή σε ποιο βαθμό βλέπουμε ότι είναι εντός περιοχής που αντιμετωπίζει γύρω-γύρω πολλές κρίσεις. Βρίσκονται αυτές οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Είναι παράγοντα σταθεροποίηση και πρέπει με αυτό το φορέα να συζητήσουμε, ώστε να καθορίσουμε ποια είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για να σταθεροποιηθεί όλη η περιοχή. Είναι προ όφελο και των χωρών της συνεργασίας, του Συμβουλίου Συνεργασία του Κόλπου και προ όφελο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Μπορούμε να συνεργαστούμε σε πολλού τομεί που θεωρεί προτεραιότητα ο φορέα αυτό και όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αναπτυχθούν. Αυτές οι χώρες είναι από τις πρώτες χώρες όσον αφορά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά ενδεχομένω ε, έχουν φανταστική δυνατότητα παραγωγής ηλιακής ε, ενέργειας ε, αυτές οι χώρες και κυρίως κατ' βουλίε των γυναικών ε, έχουν πολύ φιλόδοξη πολιτική όσον αφορά την παιδεία, την κατάρτιση και την ε, ανώτατη, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Προχωρούν γρήγορα τα πράγματα. Εδώ και κάποιο, κάποια χρόνια, 15-20 χρόνια, κάποτε, οι νέοι των χωρών αυτών έφευγαν και πήγαιναν να σπουδάσουν στη Δύση. Πήγαιναν στις Ηνωμένε Πολιτείες ή πήγαιναν στη Μεγάλη Βρετανία πιο συχνά. Σήμερα αυτές οι χώρες ακολουθούν εντελώς διαφορετική πολιτική, δεν στέλνουν πια ή τουλάχιστον και λιγότερο τους στέλνουν τους νέους τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αντιθέτως αναπτύσσουν όλες αυτές οι χώρες σημαντικότατες υποδομές στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά ζητούν συνεργασία, υπάρχουν απαιτήσει συνεργασία και όσο αφορά την κατάρτιση και την πλαισίωση του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει εκεί να είναι παρούσα η Ευρώπη και να μην αφήσει όλο αυτό το περιθώριο, αυτό το χώρο ελεύθερο για τους Αμερικανούς. Υπάρχουν μέσα εργαλεία, δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς. Παράδειγμα, για το πρόγραμμα Erasmus Mundus, οκτώ είχαμε πέρσι, μόνο οκτώ σπουδαστές που ήρθαν στην Ευρώπη σπουδαστές που προερχόταν από αυτές τις ε, αραβικές χώρες του κόλπου. Αυτές λοιπόν, αυτά τα διάφορα στοιχεία που υπογραμμίζονται στην έκθεση. Ε, προτείνω να τα συζητήσουμε τα θέματα που σκιαγράφησα. Ο κ. Ναρμπόνε, ο εκπρόσωπός μας στο Συμβούλιο συνεργασία του κόλπου στο Ριάντ είναι εδώ, παρόν, και έχω δύο ερωτήσεις να του θέσω, σύντομες. Σήμερα υπάρχουν δύο εμπόδια όσον αφορά τι διαπραγματεύσει για την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Δύο βασικά εμπόδια τέλος πάντων. Έχουμε την πολιτική ε, ρήτρα και από την άλλη πλευρά το θέμα των φόρων. Θα ήθελα να ξέρω κύριε Ναρμπόνε ε, πώς, εάν και πώς ε, θεωρείτε ότι μπορούν να υπερκεραστούν αυτά τα εμπόδια. Δεύτερον ερώτημα, κατά την άποψή σας μια τέτοια εταιρική συνεργασία πολιτική φύσεω και στρατηγική μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των χωρών του Συμβουλίου τη Συνεργασία του Κόλπου, πώ γίνονται αντιληπτά στα αίματα στι χώρε του κόλπου, τι περιμένουν αυτέ οι χώρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Αντιπροέδρε Μποντή. Αναφέρθηκε το όνομα του κύριου Ναρμπόνε και είναι και ο πρώτος που θα έπαιρνε το λόγο μετά την ε, παρέμβαση του Αντιπροέδρου κ. Μποντής. Το είχαμε σημειώσει και το δίδουμε το λόγο και τον ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχω στη συζήτησή σας. Πολύ σημαντική έκθεση αυτή για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Αν μου επιτρέψετε, θα ε, αρχίσω από το δεύτερο θέμα. Τη δεύτερη ερώτηση που έχει ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων να διανοίγονται. The ε, main thrust of the ε, Συμφωνώ με, το βασικό κορμό της έκθεσης του κυρίου Μποντής και των όσων είπε για το γεγονός ότι η περιοχή δεν γνώρισε ευξημένο ενδιαφέρον από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Το έτος 1999 ε, υπογράψα μια συμφωνία συνεργασίας και στη συνέχεια εστιάστηκα ε, το ενδιαφέρον σε τρεις ε, συμφωνίες συνεργασίας που διονύστηκαν και ακόμα δεν έχουν υπογραφεί και χρειάστηκε να επανεξετάσουμε την ανάγκη και να την επανεκτιμήσουμε για πιο στενές ε, σχέσεις με την περιοχή. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αν ενδιαφέρονται οι εταίροι μας στην περιοχή του Περσικού κόλπου ε, για μια αναθεώρηση συνολική των σχέσεων ε, και να γίνει πιο στρατηγική, βεβαίως και ενδιαφέρονται. Ε, ενδιαφέρονται πολύ ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όλη η περιοχή άλλωστε από τις αρχές του 2000 έχει αλλάξει τελείως διάθεση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπεριφορά. Είναι πιο εξωστρεφής πλέον και πολύ πιο ανοιχτή στην προσέγγιση της προς τον έξω κόσμο και ζητάει και ισχυρές σχέσεις συνεργασίας και θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, δυνητικό πρωταγωνιστή ε, στην επίλυση και περιφερειακών εκεί ε, συγκρούσεων. Θα επιθυμούσα να δείξουμε εμείς περισσότερη δέσμευση και σε πολιτικά ζητήματα της περιοχής. Ε, βεβαίως είμαστε μίζων εμπορικός εταίρος, ο πρώτος σήμερα και οικονομικός εταίρος και θεωρούν τις σχέσεις μας ως σχέσεις ε, με δυναμικό το οποίο δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί. Ε, για παράδειγμα, ε, επενδύσεις, ευρωπαϊκές εννοώ επενδύσεις στην περιφέρεια, παραμένουν χαμηλές οι επενδύσεις αυτές σε σύγκριση με άλλους εταίρους μας στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, κατανοούν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με την περιοχή και να αυξηθεί και η παρουσία της και η προβολή της εκεί. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόρπου προς το παρόν έχει στραφεί περισσότερο προς Ανατολάς, προς την Ασία και μέχρι τον Ειρηνικό και για εμπορικές σχέσεις αλλά και για επενδύσεις. Προς Ανατολάς λοιπόν ε, ε, στρέφονται και ε, περιμένουν την ανάπτυξη και του πολιτικού διαλόγου και θεωρούν, αισθάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν ναι, δεν έχει κάνει αρκετά για να διασφαλίσει τη συνέχεια στο διάλογο. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε οπωσδήποτε ότι τώρα αν θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε στη δεύτερη φάση των σχέσεών μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε πιο πολύ σε πολιτικά ζητήματα. Ναι. με πιο έντονο διάλογο και υψηλού επίπεδου. Θέλουν συνεχή λοιπόν διάλογο, ενημέρωση, ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Για θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας, το Ιράν, η σταθεροποίηση του Ιράκ, η Εμένη, ε, και θέματα Αφγανιστάν, Πακιστάν, ε, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και διάφορες άλλες περιφερειακές συγκρούσεις. Ε, βεβαίως θα ήθελαν πιο ενεργή συμμετοχή, μεγαλύτερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευρά εκπροσώπησης. Είμαστε από τις περιφέρειες που έχουμε στο ΡΙΑΤ την πιο ε, ολιγομελή εκπροσώπηση. Βέβαια είναι έξι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και υπάρχει γραμματεία. Είναι πολύ δύσκολο το έργο μας και πολύ μεγάλη δυσκολία να διατηρήσουμε πόσο μάλλον να σφυριλατούμε νέες σχέσεις όταν είναι τόσο περιορισμένη η παρουσία μας και αριθμητικά. Είναι μεγάλη η περιοχή αυτή με πολλές διαφορές. Κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της που πρέπει να μας απασχολούν και αυτές. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, βασιστούμε στα βήματα που έχουν γίνει πρόσφατα ε, με την έγκριση ενός κοινού προγράμματος δράσης για να προσπαθήσουμε επίσης να ε, κινηθούμε προς μια κατεύθυνση πιο ενεργή με μεγαλύτερη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Starting from education. Ε, αρχίζουμε λοιπόν από την εκπαίδευση. Ε, αυτή τη στιγμή ε, στη Σαουδική Αραβία είναι 60.000 οι φοιτητές τους στο εξωτερικό με πρωτοβουλίες και με υποτροφίες διμερείς όμως πάντα. Επίσης όπως είπατε ιδρύουν και νέα πανεπιστήμια γιατί αυξάνεται και ο φοιτητικό πληθυσμό. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ να αναπτύξουμε προγράμματα πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, ε, σε εταιρική σχέση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω υπάρχουν δυνατότητες όπως το Erasmus Mundus που αναφέρατε και θα ήταν ευπρόσδεκτα όλα αυτά γιατί θα αύξαναν τη δυνατότητα ε, κατάρτισης ε, δικτύων με προστιθέμενη αξία ε, πέρα από τις διμερείς σχέσεις που έχουμε έτσι κι αλλιώς. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλο το δυναμικό ε, ε, συνεργασία σε τομείς όπως είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιστήμη, τεχνολογία. Είναι πολύ βαριές οι επενδύσεις που κάνουν και ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του βασικού Κόλπου να έχουν σχέσεις και με εμάς. τους ενδιαφέρει να ανοίξουν κάποια προγράμματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις χώρες αυτές. Γιατί ε, δεν έχουμε το κλασικό μοντέλο σχέσεων εδώ του δωρητή και του δικαιούχου της ε, βοήθειας, ας πούμε. Είναι διαφορετική ποιοτικά η σχέση μας. Και το βασικό ζήτημα ή πρόβλημα δεν είναι χρηματοδότηση και δεν ενδιαφέρονται για χρήματα. Ενδιαφέρονται να έχουμε ανταλλαγές και δίκτυα και ε, σχέσεις. I uh, Τέλος, ε, θα ήταν ενδιαφέρον να κοιτάξουμε και ποια είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εντάξει, βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό πλαίσιο και το επιζητούν και εκείνοι. Ε, συζητήσαμε για εταιρικέ σχέσεις σε διάφορους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως είπα προηγουμένως, αλλά οπωσδήποτε να δούμε και ειδικά μέσα, ειδικού τρόπους ε, σύσφυξης τώρα των σχέσεων και από δική μας πλευράς, Προς το παρόν χρησιμοποιούμε το ICI ε, για πρόθεση σχετικά μικρών έργων Στο μέλλον θα χρειαστεί ίσως κάτι περισσότερο που να παίξει αν θέλετε και ρόλο καταλητικό ε, για κοινέ δράσεις, κοινέ προσπάθειες για να δείξουμε ότι είμαστε περισσότερο παρόντες. Ε, το ICI θυμίζω ότι είναι το μέσο συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες. Ε, τώρα για τις εμπορικές συμφωνίες έχουμε ζητήματα και πολιτικά και οικονομικά ε, δεν έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες εναλλαγών εδώ και πολλά χρόνια και αυτό θεωρείται, πώς να το πω, αξιολογείται αρνητικά, βαραίνει στι σχέσεις μας. Η πολιτική ρήτρα ε, για ε, το φόρο στις εξαγωγές, αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτό τον καιρό. Και ε, η θέση του Συμβουλίου συνεργασία του Περσικού Κόλπου είναι να διατηρηθεί το δικαίωμα που έχουν να επιβάλλουν φόρους στις εξαγωγές τους. Αυτό είναι κάτι όμως που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ε, καταρχήν μεν δεκτό, αλλά εντός πολλών ορίων και παραμέτρων και προϋποθέσεων και όρων. Οι συζητήσει, όπως γνωρίζετε, και οι διαπραγματεύσει έχουν οδηγηθεί σε εμπλοκή την τελευταία διετία και αυτό φυσικά δεν ε, βοηθάει στο να δημιουργηθεί θετική ατμόσφαιρα και επικοδομητική μεταξύ των δύο ενώσεων. Στο Λουξεμβούργο, στη Διευπουργική όμως ε, συνεδρίαση, θεώρησαν δύο πλευρές ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να βρούμε κοινό έδαφος και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα ή τον επόμενο μήνα συγκεκριμένα να έχουμε μεγαλύτερες και περισσότερες επαφές για να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα της επιβολής φόρων στις εξαγωγές των προϊόντων τους για να υπάρξει μια θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ναρμπόνε. Η κυρία Γιατεμάκη έχει το λόγο. Κοίτοξια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας, τον κύριο Μποντή, για την πολύ ισορροπημένη έκθεσή του και την εμπειρογνωμοσύνη του. Φυσικά εγώ δεν είμαι η Δήμων για το θέμα αυτό όπως ο κύριος εισηγητής. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να υποβάλω και κάποιες ερωτήσεις. Είναι αναφυσβήτητο ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου είναι πολύ σημαντική. Πάντως, λυπούμαστε για το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δείχνουν μεταξύ τους έναν ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τις χώρες του Περσικού κόλπου. Θα πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι, να μην έχουμε αντιπαλότητα μεταξύ μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να μιλήσουμε για την ανάγκη να είμαστε πιο συσπηρωμένοι και ενωμένοι, γιατί δυστυχώς υπάρχουν διστάμενες απόψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, καλό θα ήταν να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για την χαμηλή τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες του Περσικού κόλπου. την καλή οικονομική συνεργασία, αλλά θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε το διάλογο και να ασκήσουμε επιρροή προς χώρες αυτές, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποια θέματα κοινού ενδιαφέροντος, πολιτικά και οικονομικά και σιγά σιγά όσο θα βελτιώνεται η, η γνωριμία και η συνεννόηση μεταξύ μας να είμαστε πιο απαιτητικοί. Επίσης, σε ορισμένε επιμέρους παραγράφους. Στην παράγραφο 3, για παράδειγμα, ζητούμε να ανοίξουν νέα διπλωματικά γραφεία για να διαβριθούν οι διπλωματικές μας επαφές. Πολύ ωραία. Αλλά δεδομένη της οικονομικής κατάστασης και της ε, σοβούσας οικονομικής κρίσης και των λίγων πόρων που έχουμε, είμαστε προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να γίνει κακή χρήση των κονδύλιων εκεί. Βέβαια αυτό το ζήτημα δεν αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση του κ. Μποντής, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συνετοί, ιδιαίτερα όταν ζητούμε αύξηση της χρηματοδότησης και των πόρων. Εγώ θα προτιμούσα να επικεντρωθούμε στην αξιοποίηση των ε, υφιστάμενων πόρων και να προσπαθήσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με καλύτερη αξιοποίηση των ε, υπαρχόντων πόρων. Και φυσικά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διπλωματικών αποστολών των χωρών μελών στις χώρες του Περσικού κόλπου. Στο σημείο 5 μιλούμε για την λύπη μας ότι αφορά την απουσία ενός κεφαλαίου αφιερωμένου στον ανοιχτό, τακτικό και επικοδομητικό πολιτικό διάλογο. Γνωρίζετε κύριε εισηγητά ότι έχουμε τακτικές επαφές σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών με τις χώρες αυτές. παρόδιο αναφέρεται στο σημείο 5. Μάλιστα στο σημείο 2 προτείνεται μια στρατηγική συνεργασία, τη δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρική σχέσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Τι ακριβώς περιεχόμενο φαντάζεστε σε μια τέτοια στρατηγική εταιρική σχέση. Μήπως θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια γενική αξιολόγηση αυτών των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων. Γιατί αν έχουμε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με όλους, τότε είναι σαν να μην έχουμε κανέναν. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται κύριε Σιγητά με την πρόταση αυτή. Α, ε, δεν ήξερα αν τελειώσατε, διότι έβλεπα ότι είχατε ακόμα αναμένο το μικρόφωνο σας. Ο εισηγητής μας και ο αντιπρόεδρος ίσως ε, θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε κάποιες παρατηρήσεις και να προβεί σε κάποιο σχόλιο. πριν φύγει για τις ανελημμένες υποχρεώσεις του. κύριος Μποντής λοιπόν έχει το λόγο. <coughs> Euh, ευχαριστώ. Έχω χρόνο, μην ανησυχείτε, δεν βιάζομαι τόσο πολύ. Να απαντήσω στην κυρία Γιατερμάκη και μετά στους υπόλοιπους. Ωραία. Σας ευχαριστώ κυρία Γιατερμάκη για τα σχόλιά σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει ε, ένα ανταγωνισμό, όχι μόνο οικονομικό μεταξύ των επιχειρήσεών μα, αλλά και πολιτικό μεταξύ των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τι χώρε του Περσικού κόλπου. Και αυτέ οι αντιπαλότητε ε, ε, οι διπλωματικέ ή αυτό ο ανταγωνισμό δημιουργεί μια κακή εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Γιατί καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του νέου πλαισίου και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης να φανεί πιο σπυρωμένη, πιο ενωμένη και να ε, δίνει ένα ενιαίο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τα μέσα χρηματοδότησης και τους πόρους, θα ήθελα να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση και θα διευκρινίσω το κείμενο για να αποφευθούν τέτοιε παρεξήγησει. Εγώ δεν ζητάω αύξηση της χρηματοδότησης ε, στις χώρες του κόλπου ή αύξηση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όταν μιλώ για αύξηση των πόρων, εννοώ καλύτερη στελέχωση της αντιπροσωπείας μας εκεί. Γιατί είναι πολύ λιγομελής η ομάδα του κυρίου Ναρμπόνε στο Ριάντ. Αλλά στις πρωτεύουσε των άλλων εκει γιατι ειναι πολυ λιγο μελης η ομαδα του Συμβουλίου στις πρωτεύουσες των αλλων χωρων του Κόλπου δεν έχουμε καν αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε στο Κατάρ, ε, Ντόχα, ούτε στο Αμπουνταμπί, ούτε στο Κουβέιτ παρόλο που είναι σημαντικές ε, χώρες και σημαντικές πρωτεύουσε, δεν έχουμε εκεί καθόλου υπαλλήλου ε, αντιπροσώπους γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό είναι, χωρίς να αυξήσουμε τα κονδύλια, καλό θα είναι και σε ανθρώπινο και σε διπλωματικό επίπεδο να έχουμε καλύτερη, πιο εμφανή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όντως, εξετάζοντας την κατάσταση εκεί δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη θλίψη μας. Αν συγκρίνουμε όμως τη σημερινή κατάσταση με αυτή που επικρατούσε πριν από 10, 15, 20 χρόνια, τότε η εντύπωση είναι πιο παρήγορη. Γιατί υπάρχει μία σταδιακή προσπάθεια βελτίωσης της διακυβέρνησης στις χώρες αυτές. Υπάρχει μία βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε ανάληψη πολιτικών ευθυνών υπάρχει μια καλύτερη αναγνώριση του ρόλου των κοινοβουλίων στις χώρες αυτές. Υπάρχει μια εξέλιξη, αργή μεν, αλλά τουλάχιστον σταθερή. Δεν υπήρξαν απότομες παλινδρομήσεις, όπως ε, συμβαίνει μερικές φορές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να προβαίνει σε πολύ αυστηρές αξιολογήσεις και δρυμές αξιολογικές κρίσεις, καλύτερα να παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία που αργά αλλά σταθερά τελευταία 20 χρόνια οδεύει προς μια σωστή κατεύθυνση. Αναφερθήκατε στην στρατηγική εταιρική σχέση και εδώ συμφωνούμε ότι αν έχουμε παντού με το Μπάσα ένα εταιρική, στρατηγική εταιρική σχέση είναι σαν να μην έχουμε με κανέναν. Αλλά για την περιοχή αυτή ειδικά, για το Συμβούλιο Συνεργασία του Κόλπου, έχει νόημα αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση. Γιατί η ίδια η περιοχή είναι εξορισμού στρατηγική, έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Το Συμβούλιο συνεργασία του Κόλπου, εκτός από την Ιεμένη, εκπροσωπεί το σύνολο τη Χερσονήσου. Έχουμε την Σαουδική Αραβία και τα Αραβικά Εμμυράτα και τα Σουλτανάτα της, του Περσικού Κόλπου. Οπότε έχουμε τα στενά του Ορμούς για το κόλπο και του, τα στενά του Μπάμπελ Μαντέπ που επικοινωνεί με τον ειδικό ωκεανό και μετά μέσω του καναλιού του, Σουέ, του Σουέζ με τη Μεσόγειο Θάλασσα. Είναι στρατηγική θέση. Μην ξεχνάμε και την παρουσία της Αλκάιντα στην περιοχή. Δεν έχουμε όμως μόνο την Αλκάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέπ. Ε, έχουμε και την Αλκάιντα στην Αραβική Χερσόνησο με πολύ έντονη δραστηριότητα στην Ιεμένη. Έχουμε σχεδόν εμφύλιο πόλεμο σε, στη Βόρεια Ιεμένη. Επίσης, από τα απ την άλλη όχθη των στενών, έχουμε τη Σομαλία. Έχουμε το γειτονικό Ιράκ με την ανάγκη σταθεροποίησης αυτής της χώρας. Και απέναντι έχουμε και το Ιράν, Οπότε χρησιμοποιώ τον όρο στρατηγική εταιρική σχέση, γιατί πραγματικά η περιοχή αυτή έχει στρατηγική σημασία από γεωπολιτική άποψη, αλλά και από ενεργειακή άποψη. Γιατί αυτή η περιοχή είναι ο πρώτος μας προμηθευτής σε υδρογονάθρακες. Δεν το λέω αυτό μόνο για να φλιαρώ, δεν θέλω να κάνω λεκτικό, να προκαλέσω λεκτικό πληθωρισμό. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε ε, μία προσέγγιση προς το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου από αυτό το πρίσμα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Μιλήσαμε ε, για το θέμα του φόρου. Είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε μία απλή σχέση προμηθευτή και πελάτη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ως ένα στρατηγικό εταίρο, γιατί το θέλουμε ότι όχι, έχει αυτό το ρόλο. Θέλετε να μιλήσετε. Ναι, αλλά σύντομα παρακαλώ, γιατί πριν από το μεσημέρι έχουμε και την έκθεση του κ. Γκάλερ. Ορίστε. Ήθελα απλώς να προσθέσω κάποια πράγματα σε αυτά που ήδη ανέφερε ο εισηγητής. Ότι πράγματι αυτή είναι μια περιφέρεια, η οποία, μια περιοχή μάλλον, που έχει ισχυρούς διμερείς δεσμούς με κράτη-μέλη και όπου προφανώς υπάρχει και κάποιος ανταγωνισμός. Διότι είναι πολύ καλές αγορές ε, αναπτυσσόμενες με πολύ μεγάλο δυναμικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συμπληρωματική διάσταση αυτή σε σχέση με τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει εδώ και καιρό με κάποια κράτη-μέλη. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τέλει είναι σημαντικός εταίρος για διάφορα ζητήματα και γι' αυτό ενδιαφέρονται. Και η παρουσία μιας αντιπροσωπείας προφανώς αυξάνει την εικόνα, βελτιώνει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Θα Συζητήσουμε τις συζητήσεις και τη σχέση που είχαμε στο ΡΙΑΔ μα το, με χώρες άλλες όπου δεν υπάρχει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Και όσον αφορά τη γνώση θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσης από πλευράς των κυβερνήσεων και όσον αφορά και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί που έχουμε μια παρουσία. Αυτά ήθελα να πω για να σας δώσω μια περαιτέρω εικόνα για την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Ναρμπόνε, ε, ευχαριστώ και τον εισηγητή μας, τον κύριο Μποντής. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, να πω ότι 24 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών η συζήτηση τροπολογιών προβλέπεται για την 1η Φεβρουαρίου του 2011 και η ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 10 Φεβρουαρίου 2011 στην Ολομέλεια στη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου του 2011. Ας πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά μια βιώσιμη πολιτική Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον απότερο βορρά είναι έκθεση του κυρίου Γκάλερ που τον ευχαριστούμε που δέχτηκε να αναβληθεί η συζήτηση, να αλλάξουμε σειρά στη μερίσια διάταξη. Υπάρχουν 174 τροπολογίες που κατετέθησαν σήμερα το πρωί εντός των χρονικών ορίων. Διενεμήθη ο κατάλογος των τροπολογιών στους συναδέλφους. Το λόγο στον εισηγητή για, την ε, δύσκολο, για το δύσκολο έργο να συζητηθούν τόσες πολλές τροπολογίες. Έχετε το λόγο κύριε Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Επειδή η έκθεση κατά βάση δεν είναι επίμαχη ή αμφισβητούμενη και έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη συζήτηση και με τους γιώδης συγητές ε, στη συνέχεια ε, και διαπιστώσαμε ευρεία συνένεση. Επειδή λοιπόν συντρέχουν όλα αυτά, μπορώ να πω ευθύ εξ αρχής ότι Συμφωνώ με τις περισσότερες τροπολογίες και μπορώ να τις δεχθώ. Κατά κανόνα είναι διευκρινήσεις, συμπληρώσεις, λεπτομέρειες που στο σχέδιο της έκθεσης δεν θα είχα καν καθόλου χώρο για να τις γράψω μόνος μου, γιατί έχουμε και περιορισμούς. Γι' αυτό ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις πολύ καλές συμπληρώσεις τους. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μερικά θέματα και σε μερικούς τομείς ε, για να σας πω πού συμφωνώ να ακολουθήσουμε αυτές τις προτάσεις και πού διαφωνώ βέβαια. Ένας τομέας είναι μια ε, συνθήκη Άρκτης ε, δηλαδή για, για, την Αρκτική. Υπάρχουν τέτοιες τροπολογίες που το υπενήσονται ή το απαιτούν. Ε, δεν τις υποστηρίζω αυτές τις τροπολογίες γιατί αυτό σημαίνει ότι λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Και, ε, δηλαδή δεν μπορούμε να αποφασίσουμε χωρίς να ρωτάμε τους ενδιαφερομένους ε, και αυτό ε, προκάλεσε κάποια ενόχληση στην περιοχή ε, θορυβήθηκαν οι άνθρωποι για τις αποφάσεις αυτές που προτείνονται. Ευρύτερη μορφή συνεργασίας, καλώς. Συμφωνώ ε, με τις ε, τροπολογίες που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις δυνατότητες ε, που θα πρέπει να δημιουργούνται και να αξιοποιούνται καλώς. Τι άλλο. Στην τροπολογία υπαριθμών 20 πρέπει να σας πω κάτι γιατί στα αγγλικά λέει ενώ η βόρεια διάταξη είναι το μόνο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρηματοδοτεί την Ακτική. Δεν ισχύει αυτό αντικειμενικά. Στον προπολογισμό για την έρευνα έχουμε κονδύλια ε, από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ για το πρόγραμμα των αυριανών ωκεανών, ξέρω εγώ των θαλασσών και ε, άλλα μέσα για την Αρκτική. Αφού είμαι στη βόρεια διάσταση, εδώ στη βορειοευρωπαϊκή διάσταση, ε, πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως ε, να ασκούμε αυτή την πολιτική, την κοινή και να τη συνεχίσουμε και απέναντι στη Ρωσία, αλλά ε, η ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική δεν μπορεί να ορίζεται μέσω της βόρειο-ευρωπαϊκής διάστασης. Άλλο η Βόρεια Ευρώπη, άλλο η Αρκτική. Γιατί τα συγχαίουμε αυτά τα δύο. Κάποιος ε, μίλησε για το αρκτικό παράθυρο, Arctic Window. Μέχρι τώρα ήταν κλειστό και παγωμένο. Ε, αυτό το παράθυρο και πάντα οι Ρώσοι έλεγαν ότι εντάξει υπάρχει κάποιο παράθυρο, παράθυρο ε, όχι για πόρτα ο λόγος. Ε, ένα παραθυράκι μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να περνάμε από τη βορειοευρωπαϊκή διάσταση για να ορίζουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική. Διαφωνώ και το απορρίπτω αυτό. Στην τροπολογία 66 μια σύντομη παρέμβαση. Η συνάδελφος Γιάκον Σάρη θέλει να μιλήσει για φόρο διαχείριση των πόρων. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά ε, στην τροπολογία ε, μόνο έχει φέρει ε, μία παράθεση για τη συμφωνία μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας. Μα δεν θα το αναφέρουμε εκεί. Δεν, δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε μία συμφωνία Νορβηγίας-Ρωσίας για να βάλουμε το αηφόρο μέσα το sustainable. Άρα θα πρέπει να βρείτε να το βάλετε. Και ε, άλλες τροπολογίες ε, πολύ λεπτομερείς και πολύ εμπεριστατωμένες που αφορούν τις αρμοδιότητες των εκεί κρατών μελών. Για παράδειγμα, με ποιο τρόπο όλα αυτά μπορούν να ρυθμίζονται Παράδειγμα, η εξερεύνηση της ακτικής, ξέρω εγώ. Να σας πω ότι εννοώ συγκεκριμένα. Την τροπολογία 69 των συναδέλφων Βέσλοντ ε, και Φέρμ. Πρέπει να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε δικαιώματα εκεί ίδια. Και στην Νορβηγία, για παράδειγμα, είναι πολύ καλά ρυθμισμένα αυτά τα πράγματα με κανόνες. Δεν μπορούμε εμείς να μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες για τρίτες χώρες και να κάνουμε προτάσεις. Είμαι επιφυλακτικός. Δηλαδή, λέει εδώ, ζητάει πριν την διερεύνηση και την παραγωγή να γίνονται οι εμπειρογνωμοσύνες, να επαναεξετάζονται τα δεδομένα κτλ. Στην παράγραφο 69. Εκεί υπάρχουν αρμόδιοι φορείς, οργανισμοί που το πράττουν ήδη. Δεν χρειάζεται καμιά αναθεώρηση, reassessment, οτιδήποτε. Και είναι χώρες αυτές που έχουν οργανισμούς, υπηρεσίες, δικές τους και τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Τι δουλειά έχουμε εμεί να ανακατευόμαστε εκεί εμεί. Λες και δεν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Και η τροπολογία 70 έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα. Από πλευρά συστηματικής και μόνο δεν έχει θέση αυτό εδώ. Για το Deep Water Horizon που λέει εδώ, για την πετρελαιοκυλίδα στον κόλπο του Μεξικού. Και ε, για το πώς θα γίνεται εξόριξη και άντληση πετρελαίου στα ύδατα της Ένωσης. Ωραία, καλά είναι αυτά, αλλά ε, σε άλλη έκθεση να πάτε να το προτείνετε. Εγώ δεν κάνω λόγο στην έκθεσή μου για τα ύδατα της Ένωσης. Τι δουλειά έχει αυτό εδώ. Γι' αυτό από λόγους ε, συστηματικούς, όχι επί της ουσίας, διαφωνώ. Έρχομαι τώρα στο κλίμα. Κοιτάξτε, η Αρκτική έχει πληγεί πάρα πολύ από την κλιματική αλλαγή αλλά δεν μπορούμε εμείς με μέτρα στην Αρκτική την ίδια να αντιμετωπίσουμε ε, την κλιματική αλλαγή και να την περιορίσουμε στην ίδια την Αρκτική γιατί ε, ε, η ρήπανση δεν έχει Αρκτική ίδια. Η ατμοσφαιρική ρήπανση που επιταχύνει το λιώσιμο των πάγων και στην Αρκτική έρχεται από αλλού. Γι' αυτό χρειάζεται παγκόσμια προσέγγιση και όχι αμυγός του Βορείου Πόλου, ας πούμε, της Αρκτικής. Γιατί έρχονται από αλλού αυτά. Πάντως όλες οι δραστηριότητες ε, που, που εκτελούνται εκεί θα πρέπει να γίνονται με όσο γίνεται ε, υψηλά πρότυπα. Επαναλαμβάνω, τώρα να ζητήσουμε περιβαλλοντικά μέτρα στην Αρκτική την ίδια δεν ανατρέπουμε τίποτα ούτε περιορίζουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ε, das dazu. Ε, τώρα, έρχομαι στην τροπολογία υπαριθμών 97. Μήπως σας έχει ξεφύγει τίποτα εκεί ε, επί της ουσίας. Γιατί ζητάτε να αλλάξει ένα κείμενο με το οποίο δεν συμφωνεί η τροπολογία. Μήπως ε, καταθέσετε την τροπολογία σε λάθος σημείο. Τι έχει συμβεί ακριβώς, γιατί ζητάτε να τροποποιηθεί ένα κείμενο που δεν είναι το διπλανό. Και αυτά που, που είπαν τώρα ο Μπροκ και ο πρώην πρόεδρος δεν τα λαμβάνω καν υπόψη μου. Uh, um, λοιπόν, τι ήταν αυτή μια τεχνική υπόδειξη προς τους συντάξεις της τροπολογίας. Έρχομαι στην 103 τώρα. Η τροπολογία, για να σας τα διαβάσω στα αγγλικά, θεωρεί ε, ότι για να εντοπιστεί το ειδικό δυναμικό κάθε τόπου και να αντιμετωπιστούν και να αναπτυχθούν στρατηγικές εγκατάστασεις για διάφορες περιφέρειες με διαφορές και τα λοιπά χρειάζεται συμπερίληψη όλων και βοήθεια των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι λίγο επικουρικότητα. Εκεί πάνω εμείς δεν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δικά μας εδάφια αυτά. Τι θα πει το δυναμικό κάθε τόπου. Θα το βρει ο τόπος. Δεν θα το βρει με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δυναμικό του ο τόπος. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό και το παρακάνουμε. Καναδά, Νορβηγία, οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν και μόνοι του να τα βρουν αυτά τα πράγματα. Δεν περιμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο καλέ προθέσει και να έχουμε, το παρακάνουμε στι λεπτομέρειε. Αυτά. 112, ε, Στην 112 καλεί επιγόντως την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει ε, τα δικαιώματα, τα γλωσσικά και τα ε, πολιτισμικά των φινοουγκρικών μειονοτήτων και στη Ρωσία. Εγώ πάντα είμαι υπέρ όλων αυτών των μειονοτήτων, αλλά γιατί να το εξειδικεύουν τόσο πολύ. Στη Βόρεια Ρωσία δεν είναι μόνο οι φινοουγκρικές μειονότητες, οι άλλες να ε, υφίστανται διακριτική μεταχείριση και αυτές όχι. Όχι. Να μην επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ε, αξιοποιήσουμε τις ε, δυνατότητες που έχουμε, τις σχέσεις. Εστονία, Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, οι άνθρωποι έχουν επαφές εκεί και σχέσεις. Εμείς αυτούς να υποστηρίξουμε ε, μέσω αυτών. Αυτό είναι πιο αγνήσιο, πιο αυθεντικό. Γνωρίζουν οι ίδιοι τα πράγματα καλύτερα επί τόπου. Τώρα να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γεια σας, ήρθα να βοηθήσετε τι φιλογρικέ μειονότητε. Έχω κάνει μια τροπολογία κι εγώ που αλλάζει τη διατύπωση και νομίζω συνάδει καλύτερα με το πνεύμα των συντακτών της τροπολογίας αυτής. Αυτά. Ως προς αυτές τις τροπολογίες. Άλλες τροπολογίες τώρα υποθέτουν ή κατονομάζουν ε, ε, ε, αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της περιοχής. Κοιτάξτε, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση εδώ με την κλιματική αλλαγή γνωρίζετε ότι ανοίγουν ε, διάφορες δυνατότητες και οι ε, χώρες ε, που βρέχονται από την Αρκτική βάζουν εκεί βάσεις. Αυτό είναι και ο μόνος τρόπος έκφρασης εθνικής κυριαρχίας. Δεν είναι όλοι στρατός. Οι Rangers του Καναδά συγκρίνονται με κάποιο είδος χωροφυλακής ας πούμε στις δικές μας χώρες αστυνομία με στρατιωτική διάρθρωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει η στρατιωτικοποίηση της ακτικής. Και ε, η παρουσία των λαών του, κράτους στο ίδιο του το έδαφος δεν είναι στρατιωτικοποίηση. Ε, κάνουν αισθητή την παρουσία τους με βάση στα κράτη αυτά σε δική τους επικράτεια. Οπότε γιατί να κάνουμε τέτοιες τροπολογίες και να στέλνουμε λάθος εικόνα Αυτά. το Συμβούλιο της Αρκτικής. Κατά την άποψή μας, βεβαίως θα πρέπει να έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες εξουσίες και επιχειρησιακό να γίνει και να ε, έχει και δράση. Συμφωνούμε αλλά η διατύπωση της τροπολογίας 137 που λέει ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχυθεί το Συμβούλιο της Αρκτικής με κάθε ε, δυνατό μέσο. Και αυτό το βρίσκω λάθος προσέγγιση. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο παρατηρητές και μάλιστα ad hoc στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Οπότε δεν έχουμε και την τεράστια παρέμβαση για να ενισχύσουμε το Συμβούλιο της Αρκτικής και πάλι αυτό θα πρέπει να το θέλουν οι χώρες που είναι μέλη της Αρκτικής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ας πούμε, παρατηρητής κάθεται εκεί και βλέπει, δεν μπορεί να έχει τέτοια παρέμβαση. Βεβαίως είμαστε υπέρ ε, της ενίσχυσης, αλλά να ενισχυθεί μόνο του το Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων. Σας είπα για τη βόρειο-ευρωπαϊκή διάσταση. Ε, στην τροπολογία 142 γίνεται λόγος και πάλι για το Συμβούλιο της Αρκτικής, τη συμμετοχή των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών ενθαρρύνει το Συμβούλιο της Αρκτικής να συμπεριλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών και ΜΚΟ ως παρατηρητές ad hoc. Μα αυτό σας έχει ξεπεράσει η πραγματικότητα, ισχύει. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, διαφωνώ όμως γιατί είναι γεγονός, δεν χρειάζεται να το ζητάμε, συμβαίνει. Αυτά. Ähm, und da Έρχομαι τώρα στο πρώτο τελευταίο, ε, τροπολογία 149. Και εδώ έχω την εντύπωση λίγο ότι, πώς να το πω, πάλι είναι εκτός τόπου αυτό που ζητάνε. Το αρχικό μου κείμενο έλεγε, ή πρότεινε καλύτερα, πώς ε, θα πρέπει να οργανωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχει μια ε, συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική για την Αρκτική και τα αντίστοιχα να συμβούν και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Και ήρθε μια τροπολογία 149 που μιλάει για τελείω διαφορετικά πράγματα. Για τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν σχέση με την Αρκτική και πώς ε, θα διαμορφωθούν ε, πιο αποτελεσματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό λύστημα το θεωρώ. Κάπου αλλού μάλλον ήθελα να το υποβάλει η συντάκτρια. Ε, και το τελευταίο τώρα που θέλω να φέρω μια ενότητα θεμάτων. Όλοι οι Φιλανδοί συνάδελφοι ε, με την ίδια ακριβώ διατύπωση μου ζητούν το ίδιο πράγμα. Όχι ε, ότι με εξέπληξε και αυτό βέβαια. Ένα κέντρο ενημέρωση για την Αρκτική κέντρο πληροφόρησης καλύτερα, στο Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας. Στην έκθεσή μου το είχα βάλει λίγο πιο ουδέτερα. Και είχα πει και να υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική που να μπορεί να παρέχει βοήθεια, συνδρομή κτλ με διάβλο επικοινωνίας προς την Αρκτική από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό που ζητάτε τώρα ε, και αυτό που λέω εγώ είναι το πολιτικό μήνυμα. Πώς θα μεταφραστεί στην πράξη, πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Αυτό είναι μικροδιαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα προγράμματά της, με τα έργα της, έχει και αυτό το ρόλο να ε, συντονίζει, να οργανώνει ε, έτσι τα πράγματα ώστε να φτάνουμε στο στόχο μας. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα για τέτοιους σκοπούς, ε, ισχύουν και οι κανόνες ανάθεσης. Δηλαδή, όταν λαμβάνει κάποια μέτρα κανείς και ιδρύει ένα τέτοιο κέντρο, θα πρέπει να προκηρυχθεί και διγωνισμός με διαφόρους υποψηφίους. Έτσι είπαν αυτά. Οι κανόνες ανάθεσης έχουν κάποιες απαιτήσει. Δεν μπορώ εγώ να τα αλλάξω ή να τα προεξοφλήσω λέγοντας ότι δεν με ενδιαφέρουν οι κανόνες, εγώ θέλω να γίνει έτσι. Από πολιτική σκοπιά το καταλαβαίνω και θα το υποστήριζα, αλλά ε, θα πούνε και οι κάτοικοι της περιοχής Λαπωνίας τι ωραίο κέντρο φτιάξατε, αλλά δεν είναι το μοναδικό δίκτυο που ε, υπάρχει. Υπάρχουν και άλλα επιστημονικά που λειτουργούν πάρα πολύ καλά ήδη. Το πλήθος ε, και η πληθώρα των πληροφοριών μάλλον που φτάνουν προς τις Βρυξέλλες είναι πολύ μεγάλη. Και δεν μπορώ να, να ε, σας πω για τη διατύπωση αυτή που επιλέγετε ότι είμαι κάθετα κατηγορηματικά αντίθετος. Να βρούμε μια διατύπωση και με τους σκιώδεις που να μην χάνει το στόχο να ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε, ενημέρωση για την Αρκτική και πώς θα φτάνουν όλα αυτά στις Βρυξέλλες, αλλά και να τηρηθεί και ε, η τυπική διαδικασία που είναι απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζωή των θεσμικών οργάνων. Είμαι βέβαιος ότι στη συνεννόηση που θα έχουμε στο Στρασβούργο με τους σκιώδεις ηγητές θα βρούμε μια διατύπωση που να ικανοποιεί τους πάντες και τους Φιλανδούς συναδέλφους αλλά να σέβεται και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, ε, Αυτά. και τελειώνω εδώ την Τρίτη το πρωί την άλλη εβδομάδα στι 9 θα σα στείλω και email να έχουμε συνεδρίαση συντονιστική με του και συγκητές για να συνεννοηθούμε για να καταλήξουμε με πολύ μεγάλη συνένεση ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Το χειροκρότημα τονίζει, που την παρέμβαση συγκητή μα. Τρει έχουν ζητήσει να μιλήσουν για να σχολιάσουν. Παρακαλώ να τηρήσετε ένα τρίλεπτο καθένας διότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες μας λίγο πριν το μεσημέρι. Δεν υπάρχει άλλος αντιπρόεδρος και έχω τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου που με περιμένει. Λοιπόν, ο, καθέ, ο Σιμάνσκι και ο για τρία λεπτά. Όντω, η έκθεση αφορά ένα θέμα που δεν είναι επίμαχο, γιατί όλοι είμαστε μακριά από την Αρκτική, οπότε και οι απόψεις μας δεν είναι διστάμενες. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκάλερ, γιατί πραγματικά είναι πολύ περιεκτική η έκθεσή του, πολύ μεστή και πολύ εμπεριστατωμένη. Η Αρκτική είναι πολύ σημαντική περιοχή, αυτό είναι προφανές και Φυσικά είχαμε την πρόσφατη συμφωνία Νορβηγίας-Ρωσίας για τη θάλασσα Μπάρεντς. Είναι επικοδομητικό αυτό το, αυτή η, η συμφωνία, αλλά υπάρχουν και ανησυχητικές πτυχές όπως κάποια αφιλεγόμενα από τον Καναδά παιδεία. Οπότε υπάρχουν και θετικές και αρνητικές ενδείξεις. Εμείς στο Συμβούλιο της Αρκτικής Βρισκόμαστε σε αναζήτηση του ρόλου ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρωνόμαστε κυρίως ε, στις επιστημονικές μελέτες. Εκεί έχουμε ρόλο νομίζω να διαδραματίσουμε. Καταθέσαμε δύο τροπολογίες ότι αφορά τους νέους, τις νέες διαδρομές, τα νέα δρομολόγια. Θα πρέπει να αποφευχθούν ε, να αποφευθεί διακριτική μεταχείριση εις βάρος ορισμένων χωρών μελών σε ό,τι αφορά ε, την, τη χάραξη αυτών των ε, διαδρομών και επίσης ε, ζητήσαμε με άλλη τροπολογία τη διευθέτηση σε ό,τι αφορά τις, τις συγκρούσεις για, είτε για την υφαλοκρηπίδα είτε για τη διαχείριση των κοιτασμάτων φυσικών πόρων γιατί υπάρχουν κάποια φιλεγόμενα εκεί παιδία και κοιτάσματα που διεκδικούνται από διάφορε χώρε. Αυτά και θα καταθέσουμε τι τροπολογίε για την Ολομέλεια. Κυρία Γιάτερ Μάκη, για τρία λεπτά. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι εκτιμώ ιδιαίτερος ότι ο κύριος Πέτερνικ, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο κύριος Μπρόκο, πρώην πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, είναι και οι δύο παρόντες στη συζήτηση, επισημένοντας τον σημαντικό χαρακτήρα αυτού του θέματος. Επίση, χαίρομαι ιδιαίτερα για την πληθώρα των τροπολογιών που κατέθηκαν για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Και εγώ είμαι υπέρ ενό μόνιμου διαλόγου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των εκπροσώπων των αυτόχθων πληθυσμών ιδιαίτερα τον Σάμι. Σε ό,τι αφορά τώρα την Σκανδιναβική και τη Βόρεια Διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται στην περιοχή της Ακτικής στα πλαίσια της Βόρειας Διάστασης και η Βόρεια Διάσταση είναι μια κοινοτική πολιτική, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει και την Ισλανδία, την Ορβηγία και τη Ρωσία. Και το αρκτικό παράθυρο της βόρειας διάστασης μπορεί να χρησιμεύσει και ως ε, πρακτικό εργαλείο για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εξωτερική διάσταση του αρκτικού παραθύρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα το δυναμικό του αρκτικού παραθύρου της βόρειας διάστασης ε, δεν ε, παραμελείται από την έκθεση, το αντίθετο. Και μάλιστα συζητήθηκε και πριν από δύο εβδομάδες ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που ασχολήθηκε με τη Βόρεια Διάσταση. Και συμφωνώ και με την ανάγκη ίδρυσης ενός γραφείου πληροφοριών, ενός κέντρου πληροφοριών. Άλλωστε, οι Εστονοί συνάδελφοι συμφώνησαν με τους Φιλανδούς για την τροπολογία που αφορά το Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για το θέμα αυτό την επόμενη εβδομάδα. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερως που είχαμε την ευκαιρία που θα γίνει μια απόπειρα σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών για να συγκεράσουμε την πληθώρα αυτών των τροπολογιών. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλένσκα έχει το λόγο για τρία λεπτά. Uh, Ευχαριστώ. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση λοιπόν. Ε, και επίσης θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τον ε, ανεπίσημο χαρακτήρα του δισήματός μου. Επίσης ε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά την, τις επιστημονικές μελέτες και την παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών που είναι σημαντικά θέματα για την ε, διαμόρφωση της πολιτικής μας. Σε ό,τι αφορά το θέμα το επιστημονικό, αλλά και τα οικονομικά θέματα, γιατί η αλληλεία, η οικονομία και ο ρηκτός πλούτος αυτής της περιοχής είναι θέματα που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην, ε, οι οικονομικές αλλαγές στην περιοχή αυτή επηρεάζουν και το περιβάλλον και δεν επηρεάζουν μόνο το περιβάλλον στην Αρκτική αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και μάλιστα οι επιστημονικές μελέτες ε, στην Αρκτική δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στις χώρες που έχουν πρόσβαση στον Αρκτικό ωκεανό. Γιατί ακόμη και για τις περιοχές που καλύπτονται από διεθνείς ε, συμφωνίες και συμβάσεις, τα τελευταια δυο δύο-τρία χρόνια πολύ συχνά είχαμε υπό το πρόσχημα της ε, προστασίας του περιβάλλοντος σημαντικό περιορισμό των επιστημονικών μελετών και όχι μόνο από πλευρά της Ρωσίας. Γιατί Σίγουρα οι περιβαλλοντικέ αλλαγέ ε, στην Αρκτική και στον Οκεανό έχουν επηρεάζουν το περιβάλλον όχι μόνο στην Αρκτική ζώνη, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και οι επιστημονικέ μελέτε είναι απολύτω απαραίτητε για να κατανοήσουμε όχι μόνο τι συμβαίνει στην Αρκτική, αλλά και τι συμβαίνει και στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να περιορίζονται λοιπόν αυτέ οι επιστημονικέ μελέτε. Και δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στι χώρε που έχουν πρόσβαση στον Αρκτικό ωκεανό. Γιατί έτσι αποκλειόμαστε τελείω από το να εκφέρουμε τη γνώμη μα για τον πολικό κύκλο. Έχω καταθέσει τέσσερις τροπολογίες στην έκθεση Γκάλερ, δεν πρόκειται να τις αναλύσω, αλλά έχω κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την, το σημείο G για την αξιοποίηση των ε, φυσικών πόρων, είναι κάπω περίεργο αυτό το σημείο, γιατί δεν γίνεται αξιοποίηση αυτών των πόρων. Ίσως δεν έγινε σωστή μετάφραση αυτού του σημείου. Το πρόβλημα είναι η, αξιο... η εκμετάλλευση των ε, ζωντανών πόρων που εκεί, ε, επηρεάζουν, εκεί επηρεάζεται το κλίμα γιατί διαταράσουν το οικοσύστημα. Αυτό είναι θέμα και πολιτικό. Γιατί η γενετική πόρη, όταν λέμε μόνο γενετική πόρη και όχι ζωντανή πόρη, η γενετική πόρη είναι πολύ γενική διατύπωση και μπορούμε να περιλάβουμε τα πάντα. Ενώ όταν λέμε ζωντανοί πόροι, αναφερόμαστε στα ψάρια και στα σπονδυλωτά που χρήζουν πραγματικά ειδική προστασία. Δεύτερο θέμα. Ε, μιλούμε για Αρκτική και όχι Ανταρκτική, αλλά και ίσως ε, εκεί έγινε, ε, ήταν πρόβλημα μετάφρασης. Στο κείμενο αναφέρεται κάτι που δεν έχει επιστημονική στήριξη. Διαχείριση που στηρίζεται στο οικοσύστημα. Στη σελίδα 11, προτελευταία παράγραφος. Καλύτερα να μιλούμε για ολοκληρωμένη αξιοποίηση με σεβασμό του οικοσυστήματος. Όχι διαχείριση του οικοσυστήματος ή διαχείριση που στηρίζεται στο οικοσύστημα, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση που θα προστατεύει το οικοσύστημα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το Αρκτικό Συμβούλιο. Εκεί φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίζει την πρόταση ίδρυσης παρατηρητηρίου. Θα πρέπει να εκφράσουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της παρουσίας μας στο ε, στο Αρκτικό Συμβούλιο που θα πρέπει να είναι εκπρόσωπος από χώρες που δεν ανήκουν στο Αρκτικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και το θέμα της ίδρυσης μόνιμου παρατηρητηρίου. Στη σελίδα 15 αναφέρουν τη Δανία, η Σουηδία και η Φιλανδία. Είναι τρεις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν και στο Αρκτικό Συμβούλιο, ενώ η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το καθεστώς του μόνιμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο. Και να επανέλθω σε κάτι που είπα προηγουμένως. Δυστυχώς ήταν ε, άστοχη σε πολλά σημεία η διατύπωση εξαιτία της κακής ε, μετάφρασης που έγινε της έκθεση Γκάλερ. Καλώς, σας ευχαριστώ κύριε Βαλένσα. Τρία λεπτά και στην Επιτροπή. Είναι εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος, δεν τον ακούμε δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να πω καταρχάς ότι εκτιμούμε πολύ την πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χρειαζόμαστε προσανατολισμούς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση της αρκτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ολοκληρώνω ότι ενώ ανακοίνωση έχουμε ήδη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα συμπεράσματα του περσινού Συμβούλιου και τώρα ελπίζω πολύ σύντομα θα έχουμε και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Απότερο Βορρά. Είναι πολύ δύσκολο για μας τόσο σύντομα να αναφερθούμε στις διάφορες τροπολογίες. Ε, ίσως θα μπορούσα να σχολιάσω την διεξαχθή συζήτηση, τη σημερινή, κυρίως την παρέμβαση του εισηγητού, του κυρίου Γκάλερ. Υποστηρίζουμε σίγουρα πολλά από τα υποθέντα Κυρίω το σχόλιο ότι η βόρεια διάσταση δεν ήταν η μόνη η πηγή χρηματοδοτήσεως. Είμαστε υπερδύναμοι όσον αφορά την έρευνα που επιτρέπεται αυτό ο όρο. Και αυτό υπογραμμίζει και τονίζει αυτά που είπαν ήδη κάποιοι βουλευτές. Συμφωνούμε πάρα πολύ με το θέμα της αρμοδιότητας των διαφόρων εθνικών κρατών. Πρέπει να, προσέξουμε τα διάφορα στοιχεία της αρκτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει να προσέξουμε τα μηνύματα που στέλνουμε στις τρίτες χώρες, στους εταίρους μας στο απότερου βορρά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικότατοι όσον αφορά τη διατύπωση. Και όταν μάλιστα αναφερόμαστε στην, στα εδάφη τους, τους λαούς τους, τα ύδατά τους. Κάτι που θα ήθελα να πω άλλο είναι και το εξής. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί που αναφέρονται πράγματι θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλους τους αυτόχθονες πληθυσμού τη Αρκτική. Επίσης αληθεύει ότι οι ρωσικοί αυτόχθονες πληθυσμοί είναι κάτι που αποσχολεί περισσότερο όλου μας. Ίσως θα έπρεπε να εστιαστούμε αυτός, κυρίως στην φινογκρική οικογένεια, διότι ε, ε, ε, είμαστε κομμάτι της φινογκρικής οικογένειας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι και αυτόχθονες της φινοογγρικής ε, μειονότητας δεν θεωρούνται ως τέτοια από τη Ρωσική Ομοσπονδία και θα ήταν καλό να έχουν αυτό το καθεστώς αναγνωρισμένο από πλευράς Ρωσίας, όσοι ζουν εντός Ρωσίας. Κάτι άλλο, το Αρκτικό Συμβούλιο να είναι πιο λειτουργικό, ναι, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τη διατύπωση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο και η επιρροή μας είναι περιορισμένη. Ε, να πω κάτι άλλο. Πολλοί βουλευτές είπαν ότι είμαστε παρατηρητές ad hoc και πρέπει να συμμετέχουμε σε άλλους φορείς. Δεν υπάρχει αυτό το καθεστώς στο Αρκτικό Συμβούλιο. Όταν λέμε ότι είμαστε ad hoc παρατηρητές, τι σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται σε κάθε σύνοδο υψηλού επίπεδου κατόπιν ετήματό μας και μετά από αποδοχή των μελών, κυρίως των παρόδο και από τις ενώσεις των αυτοκτονών πληθυσμών που έχουν λόγο και θέση στο τραπέζι των συζητήσεων. Το θέμα των χρεμάτων αναφέρθηκε. Σίγουρα χρειαζόμαστε πόρους αν θέλουμε να κάνουμε πράγματα όπως βελτίωση της ε, πληροφόρησης που δίνουμε στο Αρχικό Συμβούλιο και από εσάς κατά πολύ από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τους οικονομικούς, τις οικονομικές αρχές. Ε, εσείς μας επιτρέπετε να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Η διάσταση της βόρειας διαστάσεως που αναφέρθηκε από τους βουλευτές. Ναι, θέλουμε σε κάθε ευκαιρία που συζητάμε την Αρκτική να συζητάμε το δυναμικό που έχει βόρεια διάσταση. Αλλά δεν είναι μια πολιτική στην οποία οι άλλοι μη ευρωπαϊκοί φορείς είναι παρόντες όπως ο Καναδάς, η ΙΠΑ και η Γρινλανδία. Άρα χρειάζεται να έχουμε εμείς μια δική μας ε, αρκτική πολιτική σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Γκαρσές Δελοσφάιος. Τα τελευταία τρία λεπτά ε, στον επόμενο μιλητή, τον κύριο Τάραντ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάλυψε. Ίσως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου. Ε, διότι αναφέρθηκε στους λαούς που δεν αναγνωρίζονται σε αυτόχρονες πληθυσμοί και θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Είτε είναι φινογκρικοί ε, πληθυσμοί ή με άλλη ονομασία, αλλά ζουν στην Αρκτική. Άρα είναι κάτι σημαντικό και είναι θέμα της εκθέσεως. Δεύτερο να πω ότι έχοντας την εμπειρία θητείας 18 μηνών στο Κοινοβούλιο, πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη χαρά η συνεργασία μου τον εισηγητή και τον κύριο Φαν Να κάνω μια πρόβλεψη. Μετά από δέκα χρόνια ίσως να αποκλειθούμε ως παγωθραυστικά δημιουργοί της ευρωπαϊκής ακτικής πολιτικής. Να πω στην κυρία Γιάταν Νμάκη ότι η σημερινή μας συζήτηση πυκνοκατοικείται όπως και η ίδια Αρκτική. Αλλά όλα τα σημαντικά μέλη αυτού του κοινοβουλίου είναι παρόντα, με την εξαίρεση και Χάουταλα. Προσβλέπω τη, στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, όπου έχω την εντύπωση ότι θα εξομαλύνουμε τα διάφορα προβλήματα και θα καταλήξουμε στους αναγκαίους συμβιβασμούς. Και θα προχωρήσει η έκθεση. Λοιπόν, ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Τάραντ, ήσασταν πολύ καλός, τηρήσα το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω και ο εισηγητή μας να τηρήσει τα 7 λεπτά που μπορώ να το διαθέσω για τα τελικά του σχόλια. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζομαι τόσο πολύ χρόνο, Πρόεδρε. Έτσι θα τελειώσουμε και πιο νωρί ακόμα. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων. Θέλω να πω κάτι όλους να στο συνάδελφο Βαλένσα για την έρευνα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι επιδόσεις μας και των κρατών μελών και μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο χώρος εκεί, η Νορβηγία έτσι κι αλλιώς, αλλά και ο Καναδάς ε, είναι ε, περιοχές ε, ε, πολύ αχανείς που έχουν σταθμούς ιδιωτικούς, δικούς τους, όχι ιδιωτικούς, εθνικούς, κρατικούς και συνεργάζονται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Εγώ τόλμησα να ε, εκφράσω αυτή την επιφύλαξη πρέπει να επεκταθεί, να διευρυνθεί και να το ζητάμε. Εντάξει, να δούμε πώς θα το προτείνουμε και εγώ θα υποστηρίξω κάθε αξιόλογη και αξέπαινη πρωτοβουλία σας. Πρέπει να σας πω ότι και η ρωμανική μετάφραση η γραπτή της έκθεσης δεν είναι καλή. Ε, εκμετάλλευση των γενετικών ε, ε, θαλασσίων πόρων. Τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω, τι εννοεί. να δούμε πώς θα μεταφραστεί όσο γίνεται καλύτερα. Είναι και μονοκύτταροι οργανισμοί εκεί, οι πλανκτόγκ δηλαδή που τα αλλιεύουν και τα βάζουν στη βιοτεχνολογία, στη μηχανία, αυτό εννοώ γενετική πόρη ίσως δεν είναι σωστός όρος. Θα πρέπει να δούμε αν θα μιλήσουμε για ε, Δεν ξέρω, να δω με ποιο τρόπο θα το μεταφράσουμε. Τι άλλο με ρωτήσαν. Α, ναι. Η διαχείριση με βάση το οικοσύστημα. Ε, ναι. Δυναμικό υπάρχει και εκεί θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε περισσότερο και η διατύπωση αυτή, ολοκληρωμένη διαχείριση και εμένα δεν μ' αρέσει. Θα δω... Ε, μήπως το διευκρινίσουμε καλύτερα όπως το λέτε κι εσείς. Καλώς. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα με τους και ηγητές, όπως είπα. Και θα συμπεριλάβουμε και τα όσα ακούσαμε σήμερα με τον κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Υπέροχα. Άρκεσαν τρία λεπτά για τα τελικά σχόλια. Αυτό οφείλεται στο κάποιον που ξέρει πολύ καλά ένα θέμα και μπορεί να είναι πολύ συνοπτικός και περιεκτικός. Εκτιμούμε το έργο του εισηγητού και την πλούσια σημερινή συζήτηση. Όπως γνωρίζετε, η ψηφοφορία στην Επιτροπή προβλέπεται για τις 9 Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας προβλέπεται για τις 30 Νοεμβρίου στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ σε όλους. Πέρα τη συνεδρία σα. Καλή σα μέρα.